Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, ησυχία σας παρακαλώ, διότι άρχεται η ψηφοφορία δοκιμαστικά. Καθίστε να κάνουμε μια δοκιμή σας παρακαλώ. voting cards. Παρακαλώ τις κάρτες σας να τις έχετε έτοιμες μήπως και χρειαστούν. The vote. Right. The... Right. We'll try. Right. No, mine's not working. None of them are working. Λοιπόν, δεν δουλεύει κανένα μηχάνημα. Ε, μήπως πρέπει να ανοίξετε τη ψηφοφορία. Ναι, έχουμε εδώ ένα τεχνικό σφαλματάκι. Δοκιμή παρακαλώ. Κάθεστε άνετα. Δοκιμαστικά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Καθίστε αναπαυτικά. We have 32 cards 32 κάρτες έχουμε, 27-28 ψήφισαν. Άλλοι τέσσερις παρακαλώ, 29, για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Άλλοι δύο παρακαλώ να ψηφίσουν. Ένας, άλλος κανείς. Ο αντιπρόεδρος έχει κάποια προβλήματα. Right, vote's closed and... 28 ψηφίσατε, κάθεστε άνετα, αναπαυτικά και 4 όχι. if, we, so yours doesn't work. Okay. So we have one, one extra. Λοιπόν, συν ένα ΕΛΚ παρακαλώ αν χρειαστεί γιατί δεν δουλεύει το μηχάνημα του Αντιπροέδρου σε περίπτωση που υπάρξει μικρή διαφορά. Λοιπόν, ψηφίζουμε την έκθεση του Βέρνερ Λάγκεν για τα παράγωγα, OTC και τα λοιπά. Right, we ready then? Okay. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έκθεση Λάγγεν. Έχετε όλοι τα χαρτιά σας στις λίστες σας έτοιμες. Ωραία. Τροπολογία 126, 127, 128. Μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η συμβαστική ε, AJ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η συμβαστική AK ε, στην επόμενη σελίδα. Με προφορική τροπολογία ε, των συντηρητικών. Στο τελευταίο τμήμα να προσθεθεί μία φράση. Είναι στην τροπολογία 263. Δεχόμαστε την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Προφορική τροπολογία. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική χωρίς την προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. AL στη σελίδα 5 λίγες σελίδες πιο κάτω σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το τέταρτο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα προχωρούμε στο συμβιβασμό AM, μια στιγμή να σας πω που είναι. What's this? Το βρήκαμε. Χωριστή ψηφοφορία σε 7 τμήματα. Τι συμβιβασμό είναι αν έχει 7 τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, τελικά ήταν συμβιβασμό. Και τώρα περνάμε στην συμβαστική τροπολογία AN στη σελίδα 13 λέει η πρόεδρος, εμείς έχουμε την 11 εδώ. Το βρήκατε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 393. Όχι. Καταπίπτει. 394. Ψήφι υπέρ. Η 393 καταπίπτει από ό,τι φαίνεται. Έτσι μου λένε. Η 394. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α όμικρον ο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AP με προφορική των φιλελευθέρων την οποία έχετε στα χέρια σας. Necessary, ναι, fair, reasonable. Αναγκαίο, δίκαιο και λογικό. Πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, άρα το κοινοβούλιο απορρίπτει το necessary, ναι, fair, reasonable. Καλά. Επί, χωρίς την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στο συμβασμό AQ στην επόμενη σελίδα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AR. Προσπαθώ να βρω τα δύο τμήματα και πάλι. Σελίδα 18 ή 16. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική AS. Λίγο πιο κάτω. AS υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. AT. Δύο σελίδες πιο κάτω. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AU στην ίδια σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AV στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AX στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AZ δυο σελίδες πιο κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BA πάντα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BB δεν τη βλέπω. Δεν υπάρχει συμβαστική BB, ΒΒ. Δεν έχουμε BB. I'm BB. I'm, I'm very sorry, This is, this is nothing... Συγγνώμη, Μπουρχάρτ, Μπάλτς που έχεις αρχικά BB και δεν σε έχουμε προβλέψει. Πάμε στο BC. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. BD, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν θα ψηφίσουμε την BE, αλλά πάμε στο νέο συμβιβασμό που λέγεται ZZ. <laughs> Τελικά εκεί θα καταλήξουμε, λέει ο Προεδρο. στο άρθρο 18α. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τώρα BE, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Right. BF. BF. Στην επόμενη σελίδα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. BG υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. BH υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πιο κάτω BI υπέρ, κατά, αποχές, ναι, κάντε λίγο ησυχία εκεί στη Γερμανία. Γερμανοί. BJ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. BK στην επόμενη σελίδα σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. BL. Oh, it's on the next page. All oh, right, so it is. BL in favor again. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Page BM in favor. BN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BN στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β' όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάρκου Μάρκους Φέρμπερ, τι μιλάς εκεί. Μιλάς συνέχεια, καθ' τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Δεν πειράζει. BQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BT Favor υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται BW υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. BY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο BZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CA τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται right, Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ CE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CJ υπέρ, μια στιγμή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. CK υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. CL υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. CM υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. CN υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. CO υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται CP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CY, CY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στον D τώρα. DA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DB P κατά αποχές DC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DD. Υπέρ. Oh, yeah, right. Indeed, indeed. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. 9.64 και εκτιμένη ταχύτητα. 9.64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είναι DD. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DG. Δύο προφορικές τροπολογίες. Μία των πρασίνων, πιο μακροσκελή, και μία των φιλελευθέρων που είναι συντομότερη. Με τη σειρά εμφανίσεως θα τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, την προφορική πρώτα των πρασίνων, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Των φιλελευθέρων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. Ωραία, συμβαστική DG, το αρχικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ερχόμαστε τώρα κάπου στη DH μάλλον. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα αρχίζει το αλφάβητο. Α, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Β, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Σ, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Δ, όχι, 134, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε. Okay, what fun. Compromise. Λοιπόν, συμβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 100, όχι, 152, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τη συμβαστική έτσι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική J υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική M 6 λέει εδώ όχι εδώ αν εγκριθεί η L καταπίπτει η 6 αυτό λέει εδώ συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 Υπέ κατά αποχές απορρίπτεται. 170 Υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Wow! Μπράβο Μάρκος, εσύ. 171 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική αν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Compromise O. Ε, ε, συμβαστική όμικρον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα δεν έχει σαμπάνια. 9 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται φωνή του εισηγητή. Εσείς υπέρ είστε μάλιστα εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε 182 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Ακόμα δεν έχει σαμπάνια. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα που είμαστε. Οι 2 και 185 πίπτου Συμβαστική πι. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική κιου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαμπάνια πάλι ε, συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στη 15 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 είπε. Τι λέει, καταπίπτουν. Μάλιστα, καταπίπτουν. Ο εισηγητής λέει ότι μπορούμε να ψηφίσουμε 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά υπέρ τις 214 κατά αποχές εγκρίνεται AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη όχι, διορθώνει πρόεδρος συμβαστική ΑΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Can we do this Ηλεκτρονικά παρακαλώ την τελική ψηφοφορία, το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όλα τα μηχανήματα λειτουργούν. Άλλος ένας να ψηφίσει παρακαλώ. Κλείνει. Πέρας. Εψήφισαν. 41 υπέρ, ουδής κατά και μία αποχή. Okay. Um, hang on. Μια στιγμή. Θα ψηφίσουμε και το νομοθετικό ψήφισμα. Μια στιγμή. Θέλεις το λόγο πριν ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ο εισηγητής θέλει να μιλήσει τώρα. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω ρητά όλους και να προτείνω πριν ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα, να κάνουμε μια φυσιολογικότατη πρώτη ανάγνωση τον Ιούλιο και να μην μπούμε τώρα σε διαπραγμάτευση, αλλά να έχουμε συνολική θέση του Συμβουλίου για να πάμε στη, του Κοινοβουλίου συγγνώμη, τον Ιούλιο για να πάμε στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Δεν προκάνουμε μέχρι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Και μετά να να είναι κανονική η πρώτη ανάγνωση, έτσι και αλλιώς το Συμβούλιο τσακώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια στιγμή, περιμένετε. So, so the proposal... Λοιπόν, η πρόταση είναι να, να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου πριν αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Και η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι ο συνήθως η πρόεδρος, ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές. Και η εντολή από την Ολομέλεια. Έτσι, ωραία. So does anybody want to Θέλει κανείς να πει τίποτα γι' αυτό τώρα. Συμφωνούμε όλοι. Καλώς. Ορίστε. Δύο χρόνια είμαι εδώ μέλος. Αλλά δεν είχα αυτή την εμπειρία μέχρι τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το υπόλοιπο της διαδικασίας. Yes, it means it... Σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Όχι τελική δηλαδή ψηφοφορία. Θέλεις να γίνει τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ναι. Και η τελική. Θέλεις και δεύτερη ανάγνωση. Όχι. Θέλω να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία βάση του κανονισμού και των συνθήκων να γίνει κανονική ανάγνωση στην Ολομέλεια, να ψηφίσουμε και μετά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, όχι τώρα. Να περάσει από την Ολομέλεια σε πρώτη ανάγνωση. Άρα δεν κάνουμε διαπραγματεύσει για την πρώτη ανάγνωση, θα γίνουν διαπραγματεύσει δεύτερη ανάγνωση. Έτσι λέγεται αυτό. Επίση, υπάρχει η δυνατότητα, αφού είναι πρώτη ανάγνωση, αν συμφωνήσει με όλα το Συμβούλιο, αυτά που προτείνουμε να τελειώσει ήδη από την πρώτη ανάγνωση. Αυτό που σημαίνει είναι, αυτό που λέει ο συγκητή είναι ότι θέλει να ακολουθήσει την πλήρη διαδικασία με δεύτερη ανάγνωση μετά την πρώτη. Αυτό θέλεις να, να ψηφίσουμε τώρα. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέτε αυτά. Όχι, Βίκυ, δεν μπορώ Ο, ο εισηγητής λέει θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και την τελική ψηφοφορία για να είναι θέση του, του Κοινοβουλίου. Ε, και αν δεν χτεί τη θέση του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο, πάμε σε δεύτερη ανάγνωση. Αυτό και από την αρχή. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να. Right, I'm closing the vote. Ε, κλείνει 41 υπέρ, 1 κατά και δύο εποχή. 36 υπέρ, συγγνώμη, ένας κατά και δύο εποχές. That was, that was 30... 41 σε ψήφισαν. Okay. I'm not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 παρακαλώ θέλουν να φύγουν να το πράξουν ταχαίως και όσοι συνομιλούν ιδιωτικώς να το σταματήσουν αμέσως παρακαλώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δεύτερη ψηφοφορία. Deposit Guarantee Schemes. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μια συμβιβαστική τροπολογία, συμβιβαστική 2, σε β, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, χωρίς τις λέξεις μέχρι το 10% υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα, οι, οι λέξεις μέχρι το 10% υπέρ, υπέρ, κατά, χες, απορρίπτεται. Α, όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Λέει η πρόεδρος. Δεν ήταν πάντως σαφή. Εδώ ο κατάλογος είναι λίγο μπερδεμένος. Μπερδεμένος. Είναι μακρύ το κείμενο του συμβιβασμού γι' αυτό. Τέλος πάντων, τώρα η 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νόμι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 με προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίμκο 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 13 υπέρ κατά απορρίπτεται Ήμκο 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Απορρίψες. 158 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα σι. Μακροσκελέστατη και αυτή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία του εισηγητή για την παράγραφο 3 που αλλάζει την ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι επαλήθευση για την 164 Ελέγχουμε ηλεκτρονικός την τροπολογία του Γκίγκολ 164. Έληξε. Εγκρίνεται 25 με 13. 165 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 38 τεχνική δεν ψηφίζουμε 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμκο 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική σιγματάφ F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ζήτα G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 200 έληξε απορρίφθηκε 19 υπέρ 21 κατά 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τα H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική θήτα πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που λέει investment should be in responsible υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 και 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνονται. 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 62 και οι άλλες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, μου λένε ότι 250 δεν έχει καταπέσει γιατί μιλάει για διαφορετική πτυχή του θέματος. 250 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28, ΙΜΚΟ 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, περίνεται. 64 υπέρ, κατά, Α, με συγχωρείτε. 252 πρώτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 ή πάει με τις άλλες, πάει με τις άλλες. Τότε 29 τώρα, 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμκο 29 ήταν. Ήμκο 30 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Για να το ξαναδούμε. 257 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 259 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γιώτα J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 263 υπέρ, κατά, αποχές, εγκουρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Νομική 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 265 υπέρ. Όχι, έχει καταπέσει. 266 υπέρ κατά αποχές. Για να το επαληθεύσω τη 266 πάλι. Έληξε. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 13 τζούρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές απο... Συμβιβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πηγαίνουμε στο 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2, 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστικη L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 πίπτη. 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική NM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ όχι καταπίπτει. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η Τζούρι και Ιμκο καταπίπτουν S. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 1 καταπίπτει. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χωρίς αριθμό, τι είναι αυτό. Ναι, η τροπολογία 117 με προφορική τροπολογία είναι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 118. 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 3 υπέρ, κατά, μάλλον έχει εκπέσει. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική X υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβεβαστική υψηλών Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές. Όχι δεν καταπεπτεί. Λέει πηγαίνατε στην 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ινκο 8 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 129 έχει εκπέσει. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχει καταπέσει. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα να ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες, λήξη. 34 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Yeah, I know. Do you want to do it now or later? Let's go on the resolution. Right. Then right. We'll now vote. Okay. Και τώρα... Ελάτε. Ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία ψήφους για, την, για το νομοθετικό ψήφισμα. Πέρας. 34 υπέρ, 5 κατά, μία εποχή και πάλι. Right. Right. Now, um, rapporteur. Κύριε Σεγητά. Rapporteur, we now have to, to, uh, do you Θέλετε να δηλώσετε κάτι? Θέλετε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση? Äh, Εξ όσων γνωρίζω, η Ουγγρική Προεδρία ε, στην τελευταία συνέδρια θα το συζητήσει και θα το συζητήσει αύριο. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να συμφωνήσουμε. Θα παρακαλούσα να περιμένουμε να δούμε τι στάση θα διαμορφώσει αύριο το Συμβούλιο και στο επόμενο διάστημα, εάν μπορούμε να συνεννοηθούμε και μετά να επανόλθουμε εδώ και ε, να συζητήσουμε με τους σκιώδησηγητές και στη συνέχεια να απαντήσουμε αν θέλουμε να πάμε σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση. Ε, Ωραία λοιπόν. Δευτέρα 6 Ιουνίου θα τους περιλάβουμε στην εμερήσια διάταξη για να δούμε κατά πόσον θα εγκρίνουμε εντολή για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και στις διαπραγματεύσεις της. Ε, okay, we now, we now... Και τώρα διακόπτουμε ως τις 5. Παρακαλούμε να ξανάρθετε. Θα έρθει ο Επίτροπος Μπαρνιές στις 5. Σας παρακαλώ να επιστρέψετε. Εδώ. Κυρίε και κύριοι, σφυρίζω τη λήξη του διαλύματο και μέσα τα κεφάλια. Καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Πολύ ανήσυχου σας βλέπω τέτοια ώρα. Θα ακούσουμε τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ που έχει περιορισμένο χρόνο. Όσοι ήθιστε θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις των ε, συναδέλφων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι μαζί σας για, στα πλαίσια αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου. Χθε πήγα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων άλλωστε. Αυτά τα ραντεβού για μένα είναι πολύ σημαντικά. Ελπίζω και για σας. Μπορούμε έτσι να κάνουμε έναν απολογισμό και μια αποτίμηση, ώστε να δούμε και τις προσεχείς μας συναντήσεις. Δύο διαπιστώσεις τώρα για την κατάσταση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Πρώτα απ' όλα για το ρυθμό που προχωρούν, κατά τον οποίο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Βλέπω, όπως και εσείς, ότι υπάρχει μια σχετική τόση του ενθουσιασμού και τη ε, ενεργού συμμετοχή και στην Ευρώπη και διεθνώ. Έχουμε ήδη πάρει νομοθετικά μέτρα. Η κρίση φαίνεται να βρίσκεται πίσω μα, όμω η κρίση του δημόσιου χρέου δεν έχει καμία σχέση με τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτέ οι παρατηρήσει που ακούγονται συχνά λοιπόν βρίσκονται ότι είναι επικίνδυνε. Ότι ε, αμβλύνουν την υποστήριξη τη ε, μεταρρύθμιση και ότι μπορεί να μα οδηγήσουν πάλι στο να εκτεθούμε σε υπέρμετρου κινδύνου. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αμύωτο το ρυθμό μα και αν αυτό το λέω κάπως έντονα, αυτό γίνεται γιατί η Επιτροπή είναι αποφολήτως αποφασισμένη και χρειάζεται οπωσδήποτε τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου στο έργο της. Ιδίω για να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το βασικό δίδαγμα ότι η συμπεριφορά των εμπορευομένων στο μικρό επίπεδο ε, έχει συνέπειες και στο μακροσκελέστερο επίπεδο της ε, οικονομίας. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Συστημικών Κινδύνων, που άρχισε να λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου 2011. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σημαντικό το έργο σα για το πακέτο μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση και γι' αυτό τακτικά με τεστ κοπόσεω θα παρακολουθούμε το πώ λειτουργούν τα τραπεζικά συστήματα. Συζητήσαμε στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες για αυτά τα τεστ κοπόσεως, τα συντονισμένα τεστ από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες που θα είναι πιο αυστηρά από τα προηγούμενα. Εδώ θα υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας και έντονος έλεγχος, ιδίω μέσω του συστήματος των peer reviews. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να ανασκευάζουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα μέσω από μεταρρυθμίσεις που να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση. Η δεύτερη είναι ότι υπάρχουν πολλές νομοθετικές προτάσεις μεν, πολλές ε, που επίκυνται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ετοιμάσει το σύνολο των προτάσεών της και μέσα στο, χρόνο, μέσα στο τέλος του χρόνου όλες τις υπόλοιπες, ιδίως για το τι θα γίνει μετά το G20, μετά τη συνάντηση του Λονδίνου και του Πίτσμπεργκ. Εδώ μιλάμε για ένα πακέτο νομοθετικών προτάσεων συνεπέ και συνεκτικό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, που τι παρακολουθώ πολύ στενά, διότι έχουμε συχνέ διαβουλεύσει, που από την πλευρά του ε, έχουν ενιαία διαδικασία μεταρρυθμίσεων και με, το, με τον πρόσφατο νόμο τους έχουν προβλέψει μεταρρυθμίσεις που παρόλα αυτά δεν είναι κοντά στην περάτωσή τους. Εμείς έχουμε ακολουθήσει διαδικασίες Διαφορετικέ, διότι χρειάστηκε να προβλέψουμε ένα διαφορετικό αρχιτεκτόνημα εποπτείας. Αυτό το καταρτήσαμε από κενού άλλωστε και σα καθησυχάζω εδώ, εφόσον χρειάζεται. Δεν έχω την πρόθεση να καταλήξουμε σε 20 διαφορετικές προτάσεις ε, κάθε χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Όχι κυρίες και κύριοι, τα μέτρα για την ανάπτυξη θα πρέπει προοδευτικά να αντικαταστήσουν τα μέτρα της ανασκευής. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όμως την ανασκευή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν έχουμε ξεφύγει τελείως από την κρίση. Όπως το απέδειξα και προηγουμένως, όπως φάνηκε και από τον, ε, την πράξη της ενιαία αγορά και τη στήριξη που τη δώσατε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προληπτική ή αντιδραστική ως απόκριση στην κρίση, ε, την ε, ρύθμιση λοιπόν που θα αντιμετωπίζει την κρίση, να συνεχίσουμε την ρύθμιση που θα μας επιτρέψει να περάσουμε στην ανάπτυξη. Εδώ και 1,5 χρόνο λοιπόν με τους ε, συνεργάτες μας και με αυστηρές μεθόδους παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εδώ να θυμίσω τέσσερις σημαντικές αρχές για τους προσεχείς μήνες. Πρώτον, ο συνολικός συντονισμός, ο σφαιρικός συντονισμός στο επίπεδο το διεθνές του G20 για ε, γι' αυτό το λόγο βρέθηκα πολλέ ε, μέρε στην Κίνα. Θα πάω στην ε, Ινδία και την Ιαπωνία στι αρχέ τη επόμενη χρονιά και κοιτάζουμε το Συμβούλιο Οικονομικής Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Επιτροπή της Βασιλείας και επίση ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε θα προεδρεύσω σε συνάντηση για τρει ημέρε την ερχόμενη εβδομάδα. Έπειτα θα πρέπει να έχουμε μια λεπτομεριακή βαθμονόμηση των αναγκών μα για κάθε μια από τις προτάσεις, μελετώντας και το σωρευτικό αντίκτυπο όλων των μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε απλώς να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις από τον ιδιωτικό τομέα, διότι προφανώς έτσι έχουμε εκτιμήσεις ασαφείς και γενικέ δεν λαμβάνουν πάντοτε υπόψη το γεγονό ότι οι τράπεζε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη του και να καλύψουν ένα μέρο των κεφαλαιοχικών του απαιτήσεων. Θα δημοσιεύσουμε και τι δικέ μα εκτιμήσει ταυτόχρονα με το πακέτο του υπερκεφαλαίων. Εδώ θα μελετήσουμε το μακρονομικό αντίκτυπο μια σειρά ε, οικονομικών μέτρων και θα επανέλθουμε τους ερχόμενους μήνες. Ε, ε, πλέον θα χρειαστεί μεγαλύτερο πλουραλισμό στον διάλογό μας με όλους τους συνομιλητές μας ε, για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εδώ χρειάζεται ευφυής ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων, πολύ περισσότερο από ό,τι έχει γίνει την τελευταία δεκαετία. Η δυσκολία που παρουσιάζεται είναι ότι κάποιοι όμιλοι έχουν λιγότερα μέσα από άλλου. Και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Ε, δεν μπορούν να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί. Σκέφτομαι ιδίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, τι ενώσει καταναλωτών, του αποταμιευτέ και του μικρού επενδυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, να ζητήσουμε μια νέα ισορροπία εδώ. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει δράση ώστε να έχουμε καλύτερη κάλυψη όλων των ε, ειδικών αναγκών και συμφερόντων, να ληφθούν υπόψη όλε οι απόψει, έχοντα εκπροσώπηση σε ομάδα εμπειρογνωμόνων πρώτα απ' όλα πολλοί από εσά έχετε ήδη προσκληθεί σε τέτοιε ομάδε. Ήδη έχουμε εντελεχή μελέτη τη κάθε ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, με προσοχή στη σύνθεση και τι εργασίε του. Κάτι που ήδη η γενική μα διεύθυνση το παρακολουθεί. Του ερχόμενου μήνε λοιπόν θα έχουμε σημαντική απλούστευση και αναζήτηση νέα ισορροπία στι ομάδε αυτέ, ώστε να δώσουμε περισσότερο χώρο κάτι που ε, δεν θα είναι αναγκαστικά τόσο δύσκολο στους καταναλωτές και τους υπόλοιπου συνομιλητές που αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται επαρκώ. Η γενική μα διεύθυνση στο τέλο τη χρονιά θα έχει πέντε λοιπόν ομάδε, εκ των οποίων δύο αποκλειστικώ θα ε, ε, σχηματίζονται από τι ε, κατηγορίε αυτέ που υποεκπροσωπούνται. Financial User Group και την ομάδα που θα εκπροσωπούνται οι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Έπειτα θα φροντίσουμε να δώσουμε πλήρε πληροφορίε για όλε αυτέ τι ομάδε, για την εντολή του, τη λειτουργία του στην ανάλογη σελίδα του στο τόπο της Γενικής μας Διεύθυνσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την καθοριστική έλλειψη πόρων, ώστε οι συνομιλητές αυτοί που δεν συμμετέχουν αρκετά να βρεθούν σε ισότιμη θέση με την ε, βιομηχανία, των κλάδο, κύριοι βουλευτές, έχουμε προβλέψει ένα εκατομμύριο ευρώ κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, για τον προπολογισμό του 2012 και να προβλέψουμε την ανεξάρτητη παροχή αυτή ειδική γνώση. Ιδίω στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θέλουμε να στηρίξουμε τι ενώσει που εκπροσωπούν ακριβώ του πολίτε, την κοινωνία των πολιτών. Στηρίζουμε τι ανάλογε πρωτοβουλίε, ιδίω ε, αυτά που και εσεί γνωρίζετε, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, το Financial Watch, για να έχουμε περισσότερη και εντονότερη δράση. Τέταρτη αρχή σημαντική είναι η στενότερη εταιρική σχέση με του νομοθέτε μα. Ε, του υπεύθυνου δηλαδή για την νομοθεσία. Εδώ χρειαζόμαστε συμβιβαστικέ λύσει δυναμικού χαρακτήρα. Διότι, κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εδώ θα χρειαστεί και πάλι δική σα προθυμία και ο επαγγελματισμό με τον οποίο μέσα στην ποικιλία που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο και στι πολυάριθμε κοινοβουλευτικέ σα επιτροπέ να μα κάνετε επιδομητικέ προτάσει ώστε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά που μα ενδιαφέρουν, όπω την εποπτεία, με την οδηγία IFM όλα τα θέματα που γνωρίζετε, δεν μπορώ να τα παριθμίσω τώρα, αλλά είναι σημαντικά. Και τηλεγραφικά να σας θυμίσω ότι η αρχή που θα μας καθοδηγήσει ε, στη δράση μας αφορούν πρωτοβουλίες που αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε. Οκτώ είναι τα θέματα, οι φάκελοι που σύντομα θα πρέπει να ολοκληρωθούν στην εξετασή τους. Και χωρί να περάσω στι λεπτομέρειε, απλώ να αναφέρω, ε, ευχαριστώντα εκ των προτέρων του αρμόδιου εισηγητέ των θεμάτων αυτών. Πρώτα απ' όλα, ο κανονισμό για τι πωλήσει τις ακάλυπτες. Ο εισηγητής σας έχει αναζητήσει μια γενική προσέγγιση τις τελευταίες ημέρες και το ΕΚΟΦΗΝ στις 17 Μαΐου τοποθετήθηκε ώστε τα θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν τον του διάλογο, κάτι που ξεκίνησε ήδη χθε. Θα συνεχιστούν οι σχετικέ συζητήσει. Η Επιτροπή θα διαρματίσει επίση το δικό τη ρόλο ώστε να διευκολύνει την εξέβρεση μια δυναμική λύση, όπω είπα, και εξασφαλίζοντα ένα υψηλό επίπεδο διαφάνεια για το συνολικό αποτέλεσμα διατηρώντας επίσης το δημόσιο χρέος στο επίπεδο αυτό της ρύθμισης και εξασφαλίζοντας έναν ισχυρό ρόλο στην ΕΣΜΑ λαμβάνοντα υπόψη τι μέρημνε κάποιων κρατών σχετικά με το θέμα αυτό. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα, τα παράγωγα προϊόντα και η σχετική πρόταση. Εδώ αποφανθήκατε πριν από λίγε ώρε μόλι. Πολύ σημαντικό ο κανονισμό αυτό. Πρέπει να υιοθετηθεί δυνατόν μέσα στι προθεσμίε που έχουν οριστεί, ώστε να καλύψουμε μια από τι υποχρεώσει που αναλάβαμε στο G20. Δηλαδή να προβλέψουμε υποχρεωτική αντιστάθμιση σε όλου του ε, συμμετέχοντε ε, στι αγορέ παραγόγων μέχρι το τέλο του 2012. Εδώ θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, ελπίζω σχετικά σύντομα και πάλι, τον τριμερή διάλογο. Τρίτη πρόταση, το πακέτο μέτρων Omnibus 2. Εδώ Ξέρετε ότι καλύπτεται και το θέμα της ε, solvency, solvability μάλλον 2. Ε, πρέπει εδώ να βιαστούμε, διότι θα τεθεί σε ισχύ το Solvability 2 την 1η Ιανουαρίου του 2013. Τέταρτο σημείο, οι εγγυήσει των καταθέσεων με την ε, έκθεση του κυρίου Σάιμον για την αποζημίωση των επενδυτών, επίσης του κυρίου Σμιτ. Εδώ θα πρέπει να βιαστούμε να προχωρήσουμε ακόμη γρηγορότερα να καλύψουμε και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από την υποτιμημένη τα τελευταία χρόνια άποψη που για την ώρα δεν έχει καλυφθεί. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή εδώ να δείξει ότι εντείνει τι προσπάθειε τη και να καταλήξουμε και σε ομοφωνία για το θέμα αυτό. Έπειτα οι εγγυήσει για τα ασφαλιστικά ταμεία και τι ασφαλίσει. Για το θέμα αυτό, τη σχετική πρόταση, πρέπει να πω ότι υπήρξε και η Λευκή βίβλο. δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο. Θα πρέπει την μελλοντική αυτή πρόταση να την συντονίσουμε με τι αποφάσει που θα ληφθούν για τι τραπεζικέ καταθέσει και τι αντισταθμίσεις, τι αποζημιώσεις μάλλον για τους ε, επενδυτές. Ίσως για το πέμπτο αυτό θέμα θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο παραπάνω. Και λίγα λόγια για μεγαλύτερες και κάποιες νέες, τελείως καινούργιες μεγάλες πρωτοβουλίες που θα αποσχολήσουν την Επιτροπή πέραν των όσων ήδη έχουν περάσει στο νομοθετικό πλαίσιο και στην νομοθετική του πορεία. Πρώτα απ' όλα οι νέοι κανόνες για τα τραπεζικά συστήματα. Με μια πρώτη έγκριση τα τέλη Ιουλίου. Εδώ θα υπάρξει μια οδηγία που θα περιέχει μέτρα για την εποπτεία και την συνεργασία μεταξύ των εποπτών και ένας κανονισμός ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει το κοινοτικό κεκτημένο Βασιλεία 2, τη Βασιλεία 2 και τους τεχνικούς κανόνες της Βασιλείας 3. Το θεωρήσαμε αναγκαίο αυτό για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο handbook όπως ονομάστηκε για τον τομέα αυτό. Εδώ πρέπει να χαιρετήσω και την συνεισφορά τη έκθεση Κάρα από το περασμένο Οκτώβριο, που μα φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στι διαπραγματεύσει τη Βασιλεία. Και μα ενίσχυσε στην υποβολή προτάσεων. Εδώ, σε ό,τι αφορά την ανάγκη επίση να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη Ευρώπη, και να μην ζημιώσουμε την πραγματική οικονομία ε, που χρειάζεται στήριξη και επενδύσει μακροπρόθεσμα, όλα αυτά διευκολύνθηκαν και από τη δική σα συμβολή. Δεν μπορούμε όμω σε καμία περίπτωση να μην λάβουμε αυστηρά μέτρα. Δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί, ούτε να αγνοήσουμε την απέτηση για μεταρρύθμιση. Πρέπει να δείξουμε ρεαλιστική προσέγγιση και να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη ευρωπαϊκή οικονομία και τον τραπεζικό τομέα τη Ευρώπη. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν του κανόνε τη Βασιλεία αυστηρότερα, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά στι υπόλοιπε επίρρε του πλανήτη αναγκαστικά. Τώρα, δύο άλλα σημαντικά κείμενα που πρόκειται να έχουμε σύντομα. Πρώτα απ' όλα για την αντιμετώπιση τη κρίση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε παρακολουθήσει στενά το θέμα αυτό όπως και ο κ. Φερέρα, νομίζω ότι είναι μια από τι σημαντικότερε μεταρρυθμίσει τη δική μα θητεία και τη δική μου. Δηλαδή, οι διαβουλεύσει που ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένε. Πάνω από 1.500 απαντήσει λάβαμε, ιδιαίτερη υψηλή ποιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θα λάβει υπόψη και τι συζητήσει που έγιναν με το Ευρωκοινοβούλιο και την έκθεση τη κ. Φερέιρα ε, που προανέφερα και εδώ βεβαίω θα συνεργαστούμε και με του διεθνεί μα ε, εταίρου για να εξασφαλίσουμε ένα αυστηρό επίπεδο αποτελεσματικότητα σε διεθνέ επίπεδο. Και τα μέτρα τη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να ενισχύσουν τι προσπαθίε μα. Τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση, MIFID. Για την αναθεώρηση αυτή τη οδηγία MIFID χρειάζεται να είμαστε φιλόδοξοι. Θα ακούσουμε τι απόψει όλων των ενδιαφερομένων, όχι μόνο τη Goldman Sachs ή τη JP Morgan, αλλά το σημείο κλειδί της μεταρρύθμισης αυτής θα είναι η εποπτεία όσο δυνατόν ευστοχότερη όλων των τόπων διαπραγματεύσεων και της ε, αυξημένης προστασίας και της ισότιμης ε, συναλλαγής. Έπειτα, η διακυβέρνηση των ε, επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εδώ προτείναμε μέτρα για τις τράπεζες. Αυτό είναι το τέταρτο θέμα μας. Και κάναμε συγκεκριμένε συστάσει χάρη στην έκθεση Fox που θα ληφθούν υπόψη. Οι μέτοχοι, οι αρμόδιοι σύμβουλοι και οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να έχουν συνείδηση των πράξεών τους. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Ιδιαίτερα φιλόδοξο. Ταυτόχρονα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να πάψουν τις ε, υπερβολικές υπέρμετρες αμοιβέ που είναι αδικαιολόγητε. Ε, δεν μπορούν να συνεχιστούν και δεν μπορούν και να δικαιολογούνται στο σημερινό πλαίσιο που διανύουμε. Και γενικότερα μπορώ να πω. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι επιχείρημα πλέον. Χρειάζεται χρηστή διαχείριση των κινδύνων και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ε, την αντιμετώπιση των κινδύνων με ε, σύνεση. Διότι θα πρέπει η πολιτική και ε, περιορισμένων ε, αμοιβών, αυστηρότερων, να χρησιμοποιηθεί ω τρόπο έλξη περισσότερων κεφαλαίων και να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτό το, θεωρώ, το θεωρεί αναγκαίο η Επιτροπή, γι' αυτό θα προτείνει επιπλέον μέτρα σχετικά, ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου πρακτικέ. Έχοντα βεβαίω υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει τι κανόνε παγκοσμίω στο θέμα αυτό, χωρί ε, και πραγματικά μάλλον δεν ε, φοβόμαστε ότι υπάρχει θέμα, καθώς θα συνεχίσουμε να γινώνουμε το παράδειγμα. Τώρα για τις αρχές της οδηγίας CDR3, εδώ εξετάζουμε το κατά πόσον έχει υλοποιηθεί, έχει μεταφερθεί μάλλον σωστά από ε, τα κάτι μέλη και οι διαδικασίες που παραβάσει έχουν ξεκινήσει κατά των 100 μελών που δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα μεταφοράς από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ. Κυρίε και κύριοι, προφανώ θα υπάρξουν και άλλε πρωτοβουλίε ω το τέλο τη χρονιά και με αυτά θα ολοκληρώσω. Ε, ασχολούμαστε με την τρίτη μεταρρύθμιση για του ε, οργανισμού, του οίκου μάλλον ε, αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κλίντ για την έκθεση αυτή που από την δική μα την πλευρά ήταν πάλι ιδιαίτερα χρήσιμη Μα βοηθά στο να αυξήσουμε το βαθμό διαφάνεια, για τι επενδύσει και να ασχοληθούμε με την επίλυση διαφορών, εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώ και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ποικιλία ανταγωνισμών. Αν θέλετε, σε μια αγορά που έχει συγκεντρωθεί για χύψη λόγου σε λίγα χέρια. Και ένα θέμα που μείνει ιδιαίτερα προσφυλέ, όπω και στον πρόεδρο Παρόζο, ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να αναλάβουμε δράση τη ενισχυμένη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι επενδύσει στι αναδυόμενε οικονομίε και χώρε, ιδίω για την εξορρυκτική βιομηχανία μέσω του συστηματικού reporting. Και ασχολούμαστε και με το TRIPS. Και πάλι χρειαζόμαστε κανόνε διαφάνεια και για τι επενδύσει, για τα προϊόντα, των, ε, τα επενδυτικά. Εδώ λοιπόν, Πρόεδρε, ε, θα ολοκληρώσω. Ελπίζω ότι ήμουν σαφή. Όλοι μου οι συνεργάτε ε, εργάζονται με έντονου, εντατικού ρυθμού αυτή τη στιγμή. Και Πραγματικά οι σημαντικότερε προτάσει θα έχουν φτάσει ω το τέλο του καλοκαιριού, ίσω λίγο μετά. Πάντω το πρόγραμμά μα είναι και ιδιαίτερα φιλόδοξο και χρειάζεται ενεργό συμμετοχή από όλου, ώστε να έχουμε κανόνες που να αντικατοπτρίζουν τα διδάγματα που αντιλήσαμε από την περίοδο της κρίσης, χωρίς όμως να να μειωθεί το επίπεδο επακρεπνήσής μας. Ελπίζω λοιπόν ότι με τη δική σας τη στήριξη και με τη στήριξη των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών επιτροπών θα έχουμε δυναμική ενεργό συμμετοχή εδώ, προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων για να πείσουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες που πολλές φορές με ανυπομονησία και με αγωνία και με θυμό ενίοτε περιμένουν να δουν αυτή τη διάθεση από εμάς. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές. Πρώτος ο Γκοζές και μετά οι υπόλοιποι, φιλελεύθεροι, πράσινοι κλπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν έχω ερωτήματα να σας θέσω. Γιατί περιγράψατε μπροστά μας τα πράγματα όσα έχουν και κυρίως αρχίσατε λέγοντας πολύ σοβαρά πράγματα, δηλαδή μιλήσατε για την έλλειψη θέλησης να γίνουν οι απαραίτητες ε, μεταρρυθμίσεις για τα χρηματοπιστωτικά. Αυτό νομίζω το συμμερίζονται και πολλοί από μας στο Κοινοβούλιο και της δικής μας Επιτροπής κύριο καθήκον είναι ότι η κύρια πρωτοτυπία είναι ότι πέρα από τις πολιτικές διαφορές μας προσπαθούμε να προασπίσουμε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Μιλήσατε για διάφορους συζητητές των διαφόρων ομάδων για ε, τα θέματα των οποίων εμείς καταφέραμε να συντονίσουμε τα πράγματα. Γιατί θέλουμε να υπάρξει αυτή η διευθέτηση και η επαγρύπνηση. Μερικοί νομίζουν ότι η κρίση τελείωσε, αλλά το είπατε κι εσείς, ας μην επαναλάβω ότι δεν τελείωσε ακόμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε την υποστήριξη από το Κοινοβούλιο μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών γιατί δεν ξεχάσαμε αυτά που μας είπατε όταν παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό το σέβεστε και γνωρίζουμε επίσης ότι καμιά φορά έχετε δυσκολία να το σεβαστείτε γιατί σας τίθενται εμπόδια και πολλοί σας ζητούν να το εγκαταλείψετε είπατε και σήμερα ότι δεν έχετε σκοπό να τον καταλήψετε. Εγώ ο συντονιστής βέβαια δυστυχώς επειδή δεν παίρνω πια πολλές εκθέσεις ε, θα ήθελα να σας αναφέρω μια δυσκολία μου που νομίζω θα έχει την ίδια και ο συνάδελφός μου Ούντο. Ο αριθμός των υποψηφίων για κάθε έκθεση ποιοτικών υποψηφίων έχει επιπτώσεις ως προς το ποιος αναλαμβάνει τι και μας είπατε ότι θα θέλατε να υπάρχουν κοινοί πραγματικοί, ρεαλιστικοί και αποτελεσματικοί κανόνες. Για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου που μου διέθεσε ο Πρόεδρος, θα ήθελα να σας πω απλώς ότι μπορείτε να υπολογίζετε σε εμά όπως και εμείς υπολογίζουμε σε εσά για να προχωρήσουν τα πράγματα στο θέμα αυτό. Αναφέρατε τα προσεχή προβλήματα. Το ΕΛ η ομάδα μου θα τα συζητήσει αυτά γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα του Κοινοβουλίου και γι' αυτό έχει και περισσότερες εκθέσεις αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα αναλάβουν τις εκθέσεις τους με πνεύμα συνεργασίας και του κοινού συμφέροντος. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας απογοητεύσετε με τις προτάσεις σας. Ξέρω ότι ακούγονται πολλές φήμες και από τον τύπο σε διάφορες χώρες ότι τα προσ... οι προσεχείς προτάσεις θα είναι πολύ χλιαρές και όχι αυτές που ανακοινώνονται, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή και εσείς ο ίδιος θα μας δώσετε ακριβώς τα κείμενα που χρειαζόμαστε, που να επιτρέπουν δηλαδή τη διευθέτηση των δημοσιονομικών και των χρηματοπιστωτικών. Μιλήσατε για επαλήθευση και της μεταφοράς ορισμένων τμήματων του δικαίου, όχι ως δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και επειδή είμαι και εγώ από αυτούς που συνυπέγραψαν την προηγούμενη έκκλησή σας, διαπιστώνω ότι πράγματι λάβατε υπόψη σας αυτό που ζήτησαν οι βουλευτές, δηλαδή κάποια συμμετρία στις ομάδες πίεσης, των οποίων είμαι υπέρ, γιατί μας χορηγούν πληροφορίες, δωρεάν βέβαια. Για να είναι όμως αποτελεσματικές οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να μπορούμε να έχουμε και αντιτιθέμενες πληροφορίες και απόψεις και από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει. Σε αυτά που είπατε λοιπόν κύριε Επίτροπε πρέπει να ξέρετε για αυτά που είπατε ότι σας υποστηρίζουμε. Είμαστε στο πλευρό σας ή μάλλον και μπροστά σας γιατί πολλές από αυτές τις ιδέες ε, τις πήρατε από μας. Ευχαριστούμε Ιωάννη Παύλε. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αυτόν τον καιρό όπου καθημερινά αναρωτιόμαστε εάν η Ευρωζώνη μπορεί να λύσει τα προβλήματά της, αν μπορεί να ξεπεράσει την πίεση που οργανώνουν και οι χρηματαγορές, αν μπορεί να αντέξει την πίεση αυτή και αν μπορέσουμε να δώσουμε πολιτική απάντηση που να ενισχύσει την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μήπω θα αποτύχει σε όλα αυτά η Ευρωζώνη. Για εξ ονόματο της δική μου ομάδα, θέλω να πω ότι είναι καλό που έχουμε στο πρόσωπό σας ένα συνομιλητή που μας δίνει απαντήσεις, ακούει και ε, είναι στη διάθεσή μας για συζήτηση. Καλό είναι αυτό και ωφέλιμο και βοηθάει. Και θα έχουμε να συζητήσουμε και άλλες λεπτομέρειες Γι' αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινή μας επιτυχία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο θέματα που μας καίνε κυριολεκτικά. Γιατί η κατάσταση αυτό τον καιρό επιπλέκεται και περιπλέκεται. Αφορά την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα, όμως και άλλα κράτη-μέλη και πολλά. Και όλα αυτά επιδεινώνονται από προϊόντα που δεν είναι παρκώς ρυθμισμένα και ε, από ε, πρωταγωνιστές που δεν είναι αρκετά ελεγχόμενοι και ρυθμισμένοι. Δηλαδή, όταν συζητάμε τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα ή τι μέλη γενέστε αλλού και ξαφνικά ανακύφτει το ερώτημα των CDS και πάλι, τι θα γίνει με τα CDS, πώς ρυθμίζονται αυτά νομοθετικά. Υπό την ηγεσία του συναδέλφου για το short selling έχουμε κάποια πρόοδο, αλλά το Συμβούλιο δεν βοηθάει. Διαπληκτιζόμαστε ακόμα με το Συμβούλιο γιατί δεν έχουν συμφωνήσει για τα CDS. Και αυτό είναι επισήμιο. Κοιτάξτε πώς αντιδρώνει οι χρηματαγορές και τι ζητήματα μας θέτουν και είμαστε σε θέση να επιλέξουμε το α ή το β με τα ε, credit default swaps ή χωρίς να μας επιτίθεται χρηματαγορές. Το άλλο είναι το θέμα των οίκων αξιολόγησης. Και εδώ ε, αυτοί είναι κάποιοι πρωταγωνιστές που δεν ρυθμίζονται παρκώς και το βλέπουμε αυτό. Κάποια χώρα που χρειάζεται μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές ε, και προχωρεί και σε κάποιες κινήσεις για τον προϋπολογισμό. Την παραμονή έρχεται ε, ο οίκος αξιολόγησης και ε, πατάσει την εκάστοτε κυβέρνηση με υποβαθμίσεις. Τα έχουμε συζητήσει αυτά με τον συνάδελφο Γκοζές και με άλλους σε κάποιες εκθέσεις που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί όμως. Και χρειαζόμαστε περισσότερη δέσμευση, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις έτσι ώστε πραγματικά να βγούμε από την παγίδα αυτή, την πολιτική παγίδα, εν πάση περιπτώσει, και να περάσουμε σε μια υγιή οικονομική ανάπτυξη, να επιστρέψουμε σε αυτή. Υποστηρίζουμε και εμείς εσάς και εσείς εμάς προσβλέπουμε ε, στην υποστήριξή σας. Παρακαλώ μην χαλαρώσετε τη δέσμευση γιατί είναι προϋπόθεση για την κοινή μας επιτυχία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Ούντο. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Α, και ο Φιλίπ Λαμπράξ. Μια στιγμή. Πρώτα φιλελεύθερη. Ναι, ακόμα είμαστε μεγαλύτεροι από τους πρασίνους ομάδα εδώ μέσα. Κάτι λέει ο κύριος Γκίγκολ, δεν τον ακούμε. Και εμείς λέει. Και εμείς είμαστε ακόμα μεγαλύτεροι από τους πρασίνους, λέει η κυρία Φόρτ. Εντάξει, κάντε λίγο ησυχία τώρα. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να χαιρετήσω τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ίσως να γνωρίζετε ότι δεν συμφωνώ πάντα μαζί σας, αλλά νομίζω ότι είστε ευγενέστατος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε τις απόψεις σας και θέλω να το πω αυτό. Ε, αυτά είναι εκ των όνου κάνευ. Ε, όταν συνδιαλέγεστε με πολιτικούς και όταν είστε και πολιτικός ο ίδιος, θα πρέπει να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, ακόμα και όταν δεν συμφωνούμε 100%. Θα ήθελα να πω ότι ακόμα και εγώ ως φιλελεύθερος γνωρίζω ότι θα χρειαστούμε ρύθμιση ε, σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αλλά δεν μου αρέσει ε, ο τόνος και το ύφος που χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Είναι απαραίτητο να λέμε ότι χρειαζόμαστε και το τονίζω μία ε, καλώς λειτουργούσα χρηματαγορά. Και καλές τράπεζες χρειαζόμαστε. Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά νομίζω ε, δεν τα λέμε και ορισμένοι παρακολουθούν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Και θέλω να τονίσω ότι τα προβλήματα σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα στην Ελλάδα, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι τη δικούν τη χώρα πολιτική που δεν είναι αρκετά ισχυρή. Και εγώ το λέω γιατί προέρχομαι από μια χώρα που κάναμε πολλά λάθη πριν από 15 χρόνια. Και καμιά φορά θα ήταν χρήσιμο για τους πολιτικούς αυτούς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να τις επομίζονται. Η Sharon Bowles και εγώ σας έστειλα μια επιστολή σε ό,τι αφορά ε, το σύστημα αποζημίωσης ε, της στάθμισης για τις επενδύσεις. Και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας γιατί θα το μπλοκάρουν στο Συμβούλιο και υπάρχει και ε, μειοψηφία που το μπλοκάρει. Ξέρω ότι σας ανησυχούν αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιο συμβιβασμό αν μη τι άλλο να γίνει συζήτηση πριν τις θερινές διακοπές για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Και ελπίζω να μπορέσετε να μας βοηθήσετε στην προσπάθεια αυτή. Άλλος, και συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν πολλές οδηγίες και πολλοί κανονισμοί, ε, αλλά από αυτούς ορισμένοι είναι πιο σημαντικοί για τους καταναλωτές. Κύριο Σάιμον, και το σύστημα εγγύησεως των καταθέσεων και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως ε, είναι κρίσιμα και πραγματικά κύριε Επίτροπε προσβλέπω στην υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ο Σβέν τώρα. Okay. Thank you. Um, today, as you probably... Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, σήμερα μόλις ψηφίσαμε για το ΕΜΙΡ. Και είδαμε ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει διάθεση να υπάρξει συμφωνία στην δεύτερη ανάγνωση και όχι μάλλον στην πρώτη. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο και θα δούμε αν θα υπάρξει διαπραγμάτευση ύστερα. Έχετε λοιπόν σχόλιο να κάνετε για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για το οικονομικό πλαίσιο και για το χρονοδιάγραμμα που θα ισχύσει για το όλο πακέτο. Και ιδίω πώ θα συνδυαστούμε με άλλου ρυθμιστέ διεθνώ. Από ό,τι κατάλαβα, όπω είπατε σήμερα, το MIFID, η πρόταση MIFID μπορεί να καθυστερήσει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Έτσι άφησαν να νοηθούν κάποιοι συνεργάτε σα. Για τις υποχρεώσεις σας, λοιπόν, για τα εμπορικά εργαλεία και τη διαπραγμάτευση για εμπορικά εργαλεία, δεν πρέπει να είναι όλα αυτά έτοιμα για το 2012. Ευχαριστούμε. Σβέν. Φίλιπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας να χαιρετήσω έναν μεγάλο Ευρωπαίο πολίτη παρόλο που δεν είστε του δικού μας κόμματος, ακούγοντας όμως την ομιλία σας, νομίζω ότι η πνοή που δίνετε είναι κάτι που ενδεχομένως να λείπει από κάποιους από τους συναδέλφους σας του κολεγίου. Είναι καλό λοιπόν οι επίτροποι να εκφράζονται με τρόπο φιλόδοξο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολλές φορές ακούμε ομιλίες ε, υπαναχώρησης που δύσκολα αντισταθμίζονται από άλλες φιλόδοξες ομιλίες. Για το θέμα λοιπόν αυτό το ΕΜΕΚΑΤ 4, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βιαστούμε λίγο, γιατί κάτι είπατε για τέλος Ιουνίου, φτάσαμε Ιούλιο να προγραμματίζουμε. Δεν θα είναι καινούριο για σας ότι οι κανόνες εκαθάρισης δεν θα είναι πλέον δεσμευτική ή υποχρεωτικοί. Ε, αυτό με ανησυχεί λίγο, διότι αν κάτι μάθαμε από την κρίση την οποία αντιμετωπίσαμε και τις οποίες ακόμη ζούμε τις συνέπειες σήμερα, είναι ότι το μέγιστο πρόβλημα που μα απασχόλησε και κλώνησε ιδίω στον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης ήταν η ρευστότητα. Με ανησυχεί λοιπόν πολύ το ότι μπορεί κανένα υποχρεωτικό κανόνας για το θέμα αυτό να μην ισχύει πλέον, να μην εφαρμόζεται και ιδίω για αυτή τη μεταβατική περίοδο και τις προϋποθέσεις όπου θα έπρεπε να ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο. Για μας δεν είναι αποδεκτό να επιχείρημα ότι αυτά τα, αυτοί οι μπορεί να είναι ήδη πόροι. Ενώ μπορεί κάποιες φορές ε, το μισό του κέρδος των τραπεζών να μοιράζεται σε μερίσματα και σε μπόνους. Λοιπόν, εδώ να σας θυμίσω δύο στοιχεία που δεν τα αγνοείτε σίγουρα, διότι αν και πολλές φορές έχουν ε, τύχει κακή, κακού σχολιασμού. Για, το, για τους ισότιμους κανόνες στο παιχνίδι. Ε, εδώ από κάθε άποψη, περιβαλλοντική, οικονομική, υπάρχουν ε, διεθνεί ε, προδιαγραφέ, διεθνή πρότυπα. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Το G20 δεν μπορεί να αναλάβει μια διεθνή διακυβέρνηση στα θέματα αυτά. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε αιωνίως να περιμένουμε να κινηθεί ο υπόλοιπο κόσμος για να αναλάβουμε κι εμείς δράση. Ένα δεύτερο στοιχείο η έννοια του impact assessment, τη μελέτη αντικτύπου. Το είπατε και εσεί στην προκαταρκτική στην εισαγωγή σα. Πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο των μέτρων που σχεδιάζουμε. Όμω, θα ε, είναι δυνατόν εξάντε να προβλέψουμε όλο τον αντίκτυπο όλων των νομοθετικών μέτρων που στο μέλλον θα εγκριθούν. Κανεί δεν είναι σε θέση να προβλέψει κάθε μια συνέπεια λεπτομεριακά των όσων ε, σχεδιάζονται. Ε, από οικονομική άποψη, λοιπόν, να ρωτήσω αυτού που είναι υπέρ των μελετών αντικτύπου. Πού είναι τα, τα κέρδη από τι μελέτε αντικτύπου και πού είναι οι μελέτε αντικτύπου ακριβώ για τα ζητήματα στα οποία δεν είχαν προβλεφθεί αρνητικέ συνέπειε και προέκυψαν. Λοιπόν, δεν έχουμε κανέναν που να έχει, να έχει αυτό το δικαίωμα να μα κάνει το δάσκαλο, ιδίω σε ένα κλίμα βεβαιότητα και ανασφάλεια. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα με καμία απόλυτη σιγουριά, όμω πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστούμε, Φίλιπ. Κύριε Επίτροπε, έχετε ένα σύνολο ερωτήσεων για να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο. Όχι, με συγχωρείτε. danke schön. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Ακούστηκε και προηγουμένως κύριε Μπαρνιά από εσά. Ψηφίσαμε την έκθεση Λάγκεν σήμερα και σε μία από τις αιτιολογικές σκέψεις γίνεται αναφορά ε, στην κερδοσκοπία, ε, στα τρόφιμα και τις πρώτες ύλε. Φαίνεται να γίνεται όλο και πιο καυτό αυτό το θέμα και στο γερμανικό τύπο, στο βαθμό που μπορώ εγώ να το παρακολουθήσω, γίνεται συζήτηση. Και ένα ενδιαφέρον σχόλιο είχε σήμερα η εφημερίδα Handelsblatt. Και κάποια επιμελητήρια επίσης εργατικά έχουν ε, εκφραστεί. Γίνονται δύο προτάσεις εξ όσων γνωρίζω. Η μία πρόταση είναι να αναμορφωθεί έτσι το εμπόριο ώστε να μην μπορούν οι κερδοσκόποι πλέον να έχουν πρόσβαση ε, στα χρηματιστήρια των εμπορευμάτων, ε, όχι οι κερδοσκόποι, μόνο οι έμποροι που συναλλάσσονται με τα πραγματικά προϊόντα. Ένα αυτό και δεύτερο να υπάρχει διαφάνεια ε, με νομοθετική, υποχρεωτική δήλωση όλων των συναλλαγών που γίνονται στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Και σας ερωτώ, εσείς τι φρονείτε γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέση, σε ποιο βαθμό ε, θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πριν δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο, πρέπει να σας πω ότι στην πρόταση για τους μηχανισμούς επίλυσης ε, τραπεζικών διαφορών η πρόταση θα έρθει το Σεπτέμβριο αφού θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής σε ακραίες καταστάσεις, τα περίφημα stress test. Ε, έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ε, για το σημείο αυτό κύριε Πρόεδρε, ήταν μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις για μένα κατά την εντολή μου. Να οικοδομήσουμε ένα σύστημα πρόληψης, πρόνοιας όπως λέμε στα γαλλικά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ευθύ εξ αρχή ε, στι προτάσει τη έκθεση Φεραίρα, όπω σα είπα. Ε, εδώ και καιρό, όσοι με γνωρίζουν θα ξέρουν ότι με παθιάζουν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο και την ανάληψη κινδύνου. Ε, ξέρω για, το, για όλους τους τομείς η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από ότι η επανόρθωση, η διόρθωση. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται με χρήματα που ζητάμε από τι τράπεζε για να καλύψουμε τα δικά του τα κενά και όχι από του φορολογουμένου. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια μέτρα στο κουτί των εργαλείων μα. Όμω όταν πρόκειται για την ε, πρόβλεψη, την πρόληψη. Είμαστε αρκετά έτοιμοι, αλλά δεν θα ήταν και συνετό να παρουσιάσουμε βιαστικά την πρόταση. Αυτή τη στιγμή βεβαίω έχουμε και ένα κύμα, μια σειρά από τεστ κοπόσεω. Γι' αυτό θα περιμένουμε λίγο περισσότερο μέχρι το Σεπτέμβριο για το πακέτο αυτό, το οποίο θα συνδέεται ούτω ή άλλω με όσα προετοιμάζει ο συνάδελφό μου, ο κ. Αρμούνια, για το πώ θα μεταχειριζόμαστε τι τράπεζε και από την άποψη των κρατικών βοηθειών. Εδώ λοιπόν προσπαθώ να σας περιγράψω πώς έχει συνολικά το τοπίο με δύο τέτοιες προτάσει Τη δική του για τις κρατικές βοήθειες και τη δική μας ε, για τις ε, περιπτώσεις των τραπεζών αυτές. Εδώ τώρα, κύριε Γκοζές, να πω ότι σίγουρα υπάρχει μια τάση χαλάρωσης προς την πολιτική δέσμευση, την αποφασιστικότητα εδώ, αλλά για να πω, να, να ε, θυμίσω και όσο είπε ο κύριος Μπούλμαν πριν από λίγο και για την Ελλάδα και για άλλες περιπτώσεις αυτό που οφείλουμε να κάνουμε για σκοπούς ρύθμισης, για να δείξουμε ότι αντλήσαμε τα σωστά μαθήματα από την κρίση, είναι να δώσουμε έμφαση στην εμπιστοσύνη. Να ανακτήσουμε εμπιστοσύνη, όχι πρώτα απ' όλα των αγορών, αλλά των επενδυτών, των όσων αποταμιεύουν, των πολιτών των ίδιων, την πολιτική σε εμά εμπιστοσύνη. Και μας απασχολεί ιδιαιτέρως ό,τι κάνουμε να γίνεται κατανοητό να φαίνεται ότι είναι μέτρα τα οποία μας έχουν υπαγορευτεί. Δεν με σταματήσατε στο φορολόγηση των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εδώ είμαι υπέρ στο να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία, όπως και το τι θα γίνει με τις αμοιβέ και τα μπόνους. Ναι, προτείναμε να πάμε παραπέρα, διότι θεωρούμε ότι αυτό έχει να κάνει με την ισότιμη μεταχείριση. Την, τον αγώνα που δίνουμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Κύριε Γκοζές, ε, το είπα και στην ε, Προεδρία του G20, στην κυρία Λαγκάρτ και την γαλλική κυβέρνηση, ότι εν ώψη όλων των συναντήσεων του G20 και για φέτο και για του χρόνου, προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνάντηση θα πρέπει να δούμε τι πρόοδο επιτελέστηκε σε σχέση με τι προηγούμενε συναντήσει, στο Λονδίνο, στο Πίτσπουργκ, στο, ε, στην Ουάσιγκτον, στη Σεούλ. Τι κάναμε σε σχέση με όσα μαζί αποφασίσαμε. Και εδώ για την καινοτόμα, ε, καινοτόμο ε, χρηματοδότηση, την ε, νομισματική σταθερότητα. Αυτές είναι άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσα να σας θυμίσω. Η, η διακύμανση στις τιμές των πρώτων υλών, όλα αυτά είναι θέματα σημαντικότατα. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά το πρώτο σημείο σε κάθε συνάντηση του G20 θα πρέπει να είναι πού, πώ προχωρήσαμε με τη ρύθμιση και τη διακυβέρνηση. Εάν η εξέταση αυτή γίνεται με τρόπο αντικειμενικό κάθε φορά, θα δούμε εάν υπάρχει κατά πρώτον χαλάρωση, την προσπάθεια, και έπειτα κατά πόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανησυχητικές για το τι μπορεί να γίνεται διαφορετικά από τις χώρες που κάθονται όμως στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου, κύριε Γκοζές, για το ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι μπροστά, όπως είπατε κι εσείς, αν δεν είναι στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν θα είστε πίσω μας, ως προς την ενεργό τουλάχιστον συμμετοχή σας. Αυτό το πιστεύω. Κύριε Μπούλμαν, αναφερθήκατε στην Ελλάδα, σας έχω πει την απόψή μου, για ένα από τα στοιχεία. Έπειτα υπάρχει ολόκληρο το πακέτο περί διακυβέρνησης, που με ιδιαίτερη σύνεση και επιμονή ε, σχολίαζα με τον συνάδελφο κύριο Ρεν γιατί αυτή τη στιγμή έχει μια από τις δυσκολότερες δουλειές αναλάβει και έχει και διαρκώς υποχρεώσεις εξαιτία της θέσης αυτής. Για την Ελλάδα πάντως και όλα τα θέματα που συζητήσατε και σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Κανθά για τις κάλυπτες πωλήσει. Εδώ πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Περάσαμε από το στάδιο του Συμβουλίου πριν από λίγε μέρε με μια συμφωνία που δεν ήταν και τόσο εύκολο να αποσπάσουμε, πρέπει να σα το πω αυτό, η οποία προστατεύει την πραγματική οικονομία, την πλαισιώνει όπω το είχαμε επιθυμήσει, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει και ο τριμερή διάλογο. Αυτό που μου φαίνεται εμένα ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι που δικαιολογεί την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση που δεν προέβλεπε την αυτόματη και απόλυτη απαγόρευση του short selling ή θέλαμε εδώ να δοθεί έμφαση ε, στην δυνατότητα συντονισμού των διαφορετικών εποπτών ώστε να μπορούν να λάβουν τέτοιες αποφάσεις. Αυτό το καταφέραμε να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Θα δούμε όμω πώ θα εξελιχθεί και η συζήτηση στον τριμερή διάλογο, διότι μα απασχολεί ιδιαίτερω να παραμείνει η πορεία μα φιλόδοξη. Ο κύριο Μπούλμαν έκανε ένα σχόλιο, κάτι που μου είχε πει και ο κύριο Γκοζέ για την οίκου αξιολόγηση τη πιστοληπτική ικανότητα. Ε, μα ε, απασχολεί πολύ το θέμα αυτό, η διαδικασία αποτιμησή. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνε που προβλέπει ο κανονισμό σε ό,τι αφορά την καταγραφή τις καταγραφές που ήδη έχουν ξεκινήσει, μπορούν να συνεχίσουν να βαθμολογούν εκεί, ε, εφόσον η διαδικασία καταγραφής δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν ε, έχει απορριφθεί η αίτηση για αντιδότηση. Υπάρχουν καταγραφές που από ό,τι μαθαίνω από τους συνεργάτες μου θα έχουν ολοκληρωθεί ω διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι. Κύριε Γκοζές, να σας ενημερώσω ότι κάθε οίκος ε, που έχει καταγραφεί ήδη θα μπορέσει να λειτουργήσει και στο μέλλον θα δούμε την τρίτη αναθεώρηση από το φθινόπωρο φέτος κιόλας, ώστε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην πλαισίωση και το βαθμό διαφάνειας και την ε, ποικιλία, την πολλαπλή εκπροσώπηση της αγοράς αυτής από πολλούς διαφορετικούς οίκους. Κύριε Σμιτ, να σας ευχαριστήσω για, τη, για τα καλά σας λόγια. Ναι, θέλουμε να είναι εύρωστες και σταθερές οι τράπεζες, γι' αυτό άλλωστε λαμβάνουμε νομοθετικά μέτρα όσο μπορούμε ευφιέστερα. Και χωρίς να προτρέχουμε, αλλά παραμένοντας αποφασιστικοί. Για τους επενδυτές θα πρέπει όντω να απεμπλακεί η κατάσταση στο Συμβούλιο. Η Ουγγρική Προεδρία πραγματικά δείχνει ιδιαίτερη προθυμία και μεγάλο βαθμό επαγγελματισμού, κάτι που δεν είναι και απλό για εκείνους, ε, το ανέφερα προηγουμένω. γενικώ, αλλά να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για όσα κάνει και το είπα και στην εισαγωγή μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Σμιτ, στο θέμα αυτό για την προστασία των αποζημιώσεων των επενδυτών, εδώ θα δείξουμε ε, ιδιαίτερη ευελιξία. Θα φανούμε διαλλακτικοί ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Κύριε Λαμπέρ. Με συγχωρείτε, όχι κύριε Σφέρνμπερν. Ε, αναφερθήκατε στο ΕΜΗΡ. Και η δική σας έκθεση και το πνεύμα που την συνόδευσε, ε, ναι, βεβαίως στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ε, ψηφοφορίες, τις ψηφοφορίες του, στο έργο του έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Δεν μπορώ παρά να σεβαστώ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα σας. Όμως, ε, εύχομαι να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Διότι όπως έχετε καταλάβει, οι αγορές δεν περιμένουν, τρέχουν. Πάνε πάρα πολύ γρήγορα, ιδίως αυτό το μείζον κεφάλαιο της... των παραγόγων, των παραγόγων προϊόντων. Εάν λοιπόν αποφασίσετε να περάσετε σε δεύτερη ανάγνωση, θα χρειαστούν άλλοι 6 μήνε. Έτσι δεν είναι το λιγότερο. Λοιπόν, εδώ ελπίζω να πληρωθούν οι προποθέσει. Όπω φάνηκε και σε άλλε ανάλογε περιπτώσει, με πολύ δύσκολα κείμενα, πολύ δυσκερή, όπω και το προηγούμενο φθινόπωρο μόλι, να καταλήξουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Από τη μια με την ιδιαίτερη σύνεση που σας διακρίνει από την άλλη με την ενεργό σας συμμετοχή και δεν ήταν απλό το να υπάρξει ένα αποτέλεσμα εν ώψη του G20. Αυτό είναι το γενικότερο πνεύμα που μας διέπει. Ελπίζω λοιπόν να προχωρήσετε κι εσείς σύντομα ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ενάγνωση. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Κύριε Λαμπέρ, ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. Ε, ίσως μια προσωπική παρατήρηση, ένα σχόλιο που δεν είναι άσχετο με την γενική ατμόσφαιρα που διέπει τη συζήτησή μα. Κάτι μου ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, κάτι που ακούστηκε στα λόγια σα. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότερε από τι προκλήσει και τα προβλήματα που απασχολούν και θυμώνουν του πολίτε και προκαλούν το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών χωρών είναι συνήθω διασυνοριακού χαρακτήρα, τουλάχιστον ευρωπαϊκού. Α τα δείτε ένα προ ένα, η ανάπτυξη, η ευρωζώνη, τα οικολογικά, οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση. Μπορούμε να συνεχίσουμε να τα παριθμούμε. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη απάντηση για να είναι ευστοχή θα πρέπει να έρθει από την Ευρώπη. Και έπειτα, τι βλέπουμε ταυτόχρονα. το παράδοξο που δημιουργείται είναι ότι κάθε πολιτική συζήτηση σε εθνικό επίπεδο ξαφνικά περιορίζεται. ουσιαστικά παραμένει στα στενά εθνικά όρια. Αυτό ε, δημιουργεί δυσκολίε στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και την πρόοδο. Υπάρχει απέτηση οι πολιτικοί άντρε και γυναίκε όλων των παρατάξεων, δεξιά αριστερά, ε, πράσινη, φιλελεύθερη, να δείξουν την διάθεση να δράσουν, να αποφύγουμε την επανεθνικοποίηση, την ε, την αδιαλαξία την εθνική, διότι εδώ πραγματικά καταλήγουμε σε τάσεις εθνικισμού, το τέλος της ε, ενιαίας αγοράς που είναι η βάση της ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τα λέω αυτά ίσως κάποιος έντονα, αλλά με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό και ισχύει και για τα οικονομικά ζητήματα που μας απασχολούν. Για το CDR4 και την ρευστότητα. Κύριε Λάμπερτ, θα υπάρξουν κανόνες γενικοί για την ρευστότητα στην πρότασή μας. Γιατί σε κάθε περίπτωση προτίθεμαι να λάβω υπόψη τις συστάσεις της Βασιλείας ώστε να υλοποιηθούν και στην πράξη, στην πραγματική οικονομία όλα όσα προβλέπονται εκεί. Θα λάβουμε λοιπόν διατάξει σχετικά με τη ρευστότητα και θα προβλέψουμε αυστηρού κανόνε για όλε τι τράπεζε. Θα πρέπει να διαθέτουν διαρκώ την... τα απαραίτητα αποθέματα ρευστού. Και αυτό θα πρέπει να μπορούν να το παρακολουθούν και οι επόπτε. Τα... Κατά τα άλλα, σα επισημαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικώ ιδιαίτερα περίπλοκο, με σοβαρού αντικτύπου στην στην πραγματική λειτουργία τη οικονομία. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι εκεί στην ίδια τη Βασιλεία προβλέφθηκε αυτός τα πλαίσια της ε, Γενικής Συμφωνίας. Θα κάνουμε λοιπόν ένα, μια πραγματική προσπάθεια για τις ε, πραγματικές αναλογίες εφόσον ολοκληρωθεί η προσπάθεια αξιολόγησης, βαθμονόμησης εφόσον να βρεθούν αυτά τα νέα σημεία ισορροπία, ώστε να έχουμε πολύ ακριβεί αναλογέ, πολύ ακριβή ποσοστά. Εδώ λοιπόν παρακολουθώ το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. Διατηρώ την φιλοδοξία να προστατεύσουμε την πραγματική οικονομία και να σεβαστούμε και όλους τους κανόνες της Βασιλείας, όμως να μην ξεχάσουμε ότι είναι δύο φορές ε, ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης σε σχέση με όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Δηλαδή από τη μια τα τρία τέταρτα τη ε, ευρωπαϊκή οικονομία χρηματοδοτούνται από τι τράπεζε και όχι το ένα τέταρτο όπω στι ΗΠΑ, τα τρία τέταρτα. Και εμεί επιλέξαμε να εφαρμόζουμε του κανόνε τη Βασιλεία σε όλε τι τράπεζε. Όχι μόνο σε 15-20. Εάν εφαρμόζαμε του κανόνε τη Βασιλεία όπω κάνουν οι Αμερικανοί στι μεγαλύτερε μόνο ευρωπαϊκέ τράπεζε, θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Αλλά εμεί αποφασίσαμε να ισχύουν αδιακρίτω για όλε τι τράπεζε ε, τα ε, οι αυτοί. Αυτό κάνει, μας δίνει 8.000 τράπεζες στην Ευρώπη. Ο κύριος Λάμπερτς ανέφερε τον ε, σωρευτικό αντίκτυπο αυτών των μεταρρυθμίσεων και των σχετικών αναλύσεων. Πρέπει να αναρωτηθούμε εάν ο κλάδος αυτός είναι ο ίδιος ε, στην καλύτερη θέση ώστε να, ο ίδιος να αποτιμά τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές του. Μα προφανώς ε, υπάρχουν μελέτες αντικτύπου που πολλές φορές δημοσιεύονται με τρόπο πολύ Αλλά εδώ κάποιες φορές ε, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος, ούτε και το όφελος που θα εκπροσωπούσαν τέτοιε μελέτε εφόσον γίνονται σωστά για μα, δηλαδή τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Εδώ τώρα το Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Σχέσεων. Ω παράδειγμα το λέω αυτό, όρισε ότι το ΑΕΠ τη Ευρωζώνη μπορεί να μειωθεί ω το 2014 κατά 4,7% αν εφαρμόσουμε πιστάλλου του κανόνε τη Βασιλεία 3. 4,7%. Και η Επιτροπή της Βασιλείας ταυτόχρονα εκτιμά ότι ο αντίκτυπος θα είναι πολύ υπιότερος. Εκτιμώντα ότι το διεθνές ΕΕ μπορεί να μειωθεί κατά 0,19%. 4,5% μετά την θέση σε ισχύ βασιλείας. Βασιλεία. Εδώ ο καθένα βέβαια μπορεί να πάρει και να κρατήσει ό,τι θέλει από όλα αυτά ακούει όλες τις απόψεις και μπορεί να συγκεντρώσει τις μελέτες αντικτύπου όλων και να αποφασίσει τι μπορεί να ισχύει. Εδώ σε αυτό που αναφερθήκατε και το οποίο μας απασχολεί εδώ και καιρό, να σας διαβεβαιώσω ότι, κύριε Κουτέ, κύριε Κλούτε, για την αγορά παραγόγων και τι πρώτε ύλε, Το θέμα αυτό μα απασχολεί εδώ και καιρό, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Η διακύμανση των τιμών, που είναι πολύ έντονη μάλιστα σε ορισμένε χώρε, ιδίω στι αφρικανικέ χώρε που γνωρίζω καλά, η εξάρτησή του από τι εξαγωγέ τροφίμων πολλέ φορέ φτάνει το 40%. Οι διακυμάνσει λοιπόν στις τιμές πλήττει, για να μην πω, κάνει τις χώρες αυτές να ασφικτιούν το κόστος μόνο για τη Σενεγάλη από ρύζι Ταϊλάνδης φτάνει 2-3 μονάδες του ΑΕΠ για μια χώρα που έχει ένα ποτάμι μεγάλο που διασχίζει τη χώρα με πολύ νερό έτσι θα μπορούσε να υπάρχει αγροτική καλλιέργεια πολύ οργανωμένη και να μειωθεί και να περιοριστεί Σοβαρά η εξάρτηση αυτή. Το πρώτο, λοιπόν, η πρώτη συνέπεια από τις διακυμάνσεις των τιμών, κύριε Κλούτε, είναι στην ισορροπία ε, προσφοράς και ζήτησης σε μια περίοδο που για διαφορετικούς λόγους η προσφορά βρίσκεται σε τέλμα, τουλάχιστον δεν αυξάνεται. Από τη μια έχουμε πλημμύρε, από την άλλη ε, λειψιδρία, από την άλλη κλιματικά ακραία φαινόμενα. Και η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται, δεν θα πάψει να αυξάνεται. Μην ξεχνάμε ότι κατά 50% έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, έχει διπλασιαστεί μάλλον, η αγροτική παραγωγή. Θα πρέπει να διπλασιαστεί μάλλον η αγροτική παραγωγή αν θέλουμε να καλύψουμε τα 9 δις, 9 δις του ανθρώπινου πληθυσμού στο 2040. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι η ε, οικονομική αστάθεια και έπειτα τα όσα προκαλεί η κερδοσκοπία. Η αστάθεια και η βεβαιότητα προκαλούνται από την κερδοσκοπία. Σε δύο λοιπόν επίπεδα πρέπει να δράσουμε. Πρώτα απ' όλα στη διαφάνεια, όπου προσπαθώ να συμβάλλω όσο γίνεται περισσότερο ίδια με τα παράγωγα προϊόντα, να δούμε τι κάνει ο καθένα και ο καθένα βέβαια να υποχρεώται να αναλάβει τι ευθύνε του. Όταν ε, η κερδοσκοπία ξεπερνά κάποια όρια, θα πρέπει να υπάρχουν ε, και οι ανάλογε κυρώσει. Και στα ανάλογα ευρωπαϊκά κείμενα πρέπει να πλαισιώνονται οι διάφορε θέσει. Αν δεν θέλουμε ο ίδιος παράγοντας, ο ένας και μόνος να κυριαρχήσει όλη την αγορά και να στρεβλώσει ολόκληρο τον ανταγωνισμό. Τότε όπως και οι Αμερικανοί πρέπει και εμείς στο μυθείο να προτείνουμε περιορισμούς, όρια. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ναι, ε, εγώ είμαι πρεσβύτερο μέλος, γι' αυτό προεδρεύω, γιατί δεν υπάρχει άλλος αντιπρόεδρος εδώ να προεδρεύσει. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, στη συζήτηση. Κυρία Μακάρτη πρέπει να φύγει, γι' αυτό θα μιλήσει πρώτη. Είναι με έναν αντιπρόεδρος, αλλά πρέπει να φύγει, γι' αυτό δεν προεδρεύει εκείνη. Ναι, έχω ανηλυμένη υποχρέωση μία ραδιοφωνική συνέντευξη με τους εκλογείς μου. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στα σχόλια του κυρίου Γκοζές, δηλαδή πρέπει πόντος να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση που προτείνεται κύριε Επίτροπε και όπως είπε και ο κύριος Σμιτ θέλουμε επίσης να υπάρχουν υπεύθυνε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χωρίς να αυτορυθμίζονται μόνες τους. Σε μερικά από τα blog και τα άρθρα που διαβάζω στο ίντερνετ για την αγορά των credit default swaps βλέπω φράσεις όπου λένε εμείς ως πολιτικοί δεν θέλουμε να γίνει κυνήγι μαγισσών, δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τις τράπεζες και τις έρευνες τις κάνουμε μόνο γιατί υπήρξαν κακές δημόσιες σχέσεις. Πράγμα που δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί λένε σε αυτά τα άρθρα δεν παίρνουν στα σοβαρά το ρόλο τους και δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να μην δίνεται η εντύπωση ότι ό,τι λέμε το κάνουμε απλώς και μόνο για να στηρίξουμε τα συμφέροντα των τραπεζών. Ένα ερώτημα κύριε Επίτροπε. Δουλειά μας είναι η νομοθεσία, αλλά επίσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής ή μη της νομοθεσίας. Και πολλοί συνάδελφοι πρόσεξαν ότι στη δική μου έκθεση πολλές χώρες μέλη εφαρμόζουν τη μεταρρύθμιση, όχι μόνο μία, αλλά την εφαρμόζουν όπως θεωρούν σωστό και μάλιστα σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Όλε οι χώρες μέλη συνυπέγραψαν τη συμφωνία αλλά την, ερμηνεύει κάθε μία χωριστά, διαφορετικά. Η Κομισιόν λοιπόν δεν θα μπορούσε από κοινού με το Κοινοβούλιο, το προσωπικό και τους βουλευτές να οργανώσει μία ακρόαση, ένα τεχνικό εργαστήριο για να δούμε γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά μεταξύ της νομοθεσίας και της εφαρμογής της διότι νομίζω ότι πρόκειται για θέμα που δημιουργεί προηγούμενο για κάθε νομοθέτημα, όχι μόνο για αυτό για τη χρηματοπιστωτικά. Επίσης, επειδή μερικοί από εμά πηγαίνουν σήμερα στην Ιρλανδία για να συζητήσουν ακριβώς εκεί την κρίση, σε τι βαθμό ψάχνετε εναλλακτικέ λύσεις για το πρόβλημα, γιατί όπως και να το δούμε η κατάσταση στην Ιρλανδία δεν είναι ε, ικανοποιητική και ούτε βελτιώνεται και οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος σε ύψος 50.000 ευρώ κατά κεφαλήν μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την επιβάρυνση του φορολογούμενου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί νομίζω μια, μια, ένας δρόμος όπου η, την κρίση να αντιμετωπίζουμε με ταχύτητα που δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Χαίρομαι που θα πάτε στην Ουάσιγκτον και γενικότερα στις ΗΠΑ για να δείτε τι γίνεται για τη μεταρρύθμιση εκεί των χρηματοπιστωτικών παγκοσμίω. Γι' αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω την επόμενη φορά που θα πάτε και θα συναντήσετε το Γενικό Εισαγγελέα εκεί που έχει αναλάβει μία έρευνα για το ρόλο ορισμένων τραπεζών στην κρίση να με ρωτήσετε μήπως δεν θα έπρεπε και εμείς να εξετάσουμε το ρόλο που έπαιξαν οι τράπεζες στην κρίση ας πούμε για την κρίση στην Ιρλανδία γιατί πολλοί πιστεύουν ότι φταίνε οι κυβερνήσεις και όχι οι τράπεζες και οι ίδιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Έχουμε ακόμα 7 ομιλητές. Θα σας παρακαλούσα να μην μακρηγορείτε τόσο πολύ όσο η αντιπρόεδρος μας. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γκίγκολτ. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, ο συνάδελφός μου Φιλίπ ε, είπε ποια είναι η δική μας άποψη και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Γνωρίζετε ότι συμφωνώ. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ποια είναι η ησυχία μου αυτό τον καιρό. Μπορεί να είδατε τις διαμαρτυρίες στην Ισπανία με σύνθημα πραγματική δημοκρατία. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτά. Είδαμε ε, τώρα ε, τις πρώτες διαμαρτυρίες στην ε, πλατεία Βαστήλης του Παρισιού και στην πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Και στην Ιρλανδία ο κόσμος διαμαρτύρεται και ουσιαστικά όλοι λένε ότι το κόστος αυτής της κρίσης δεν θα πρέπει να το πληρώσει ο κόσμος. Δεν το πληρώνουν οι υπεύθυνοι, δεν προχωράει ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Ξέρω ότι έχετε αντίθετη άποψη και δεν συμφωνείτε, έχει βλοκάρει αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι οι πιο αδύναμες χώρες επιβαρύνονται όλο και περισσότερο, ενώ οι πιο ε, πλούσιες χώρες από την οποία και εγώ προέρχομαι θεωρούν ότι είναι εντάξει και ότι ήταν ανέκαθεν εντάξει τα πράγματα. Οι ισχυρέ χώρες στην Ευρώπη όμως δεν μπορούν να λύσουν την κρίση και χάνουμε ε, ακριβώς την αιτία. Τι έγινε, ότι κάποιες αγορές επένδυσαν σε λάθος ε, τομείς. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και ε, ο ιδιωτικό τομέας, βέβαια έφτυγε και το κράτος γιατί είχε λάθο κανόνες και ρυθμίσεις. Και τώρα ε, διαβλέπω τον εξή κίνδυνο και απευθύνομαι σε εσά. Γιατί ξέρω ότι σκέφτεστε το θέμα των χρηματαγορών όχι μόνο τεχνικά αλλά και πολιτικά. Γνωρίζουμε ότι μειώνονται οι απαιτήσει ρευστότητα ε, στους κανόνες της Βασιλείας κατά την εφαρμογή τους. Επίσης, βλέπω σε κάποια έγγραφα ότι δεν θέλετε ε, δίκτυ μόχλευσης, ε, leverage ratio, αλλά στα stress test δεν έχουν καταφέρει ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι εποπτικές αρχές να βρουν αξιόπιστα τεστ. Το έχουν πει όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ρωτήσαμε και δεν μας απαντούν γιατί δεν γίνονται αυτά με τρόπο σωστό και ε, τι γίνεται με τα ρίσκα των δημοσίων δανείων και για να το πω έτσι με όρους πολιτικούς. Εάν εσείς, ε, τελειώνω σχεδόν, για να το πω λοιπόν σαφώς και σύντομα, εάν δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει χώρο στα λόμπι να βάλουν τις εξαιρέσεις στους κανόνες ε, για να μην είναι συνεπείς στη ρύθμιση των χρηματαγορών και στη γρήγορη εφαρμογή των προτάσεων για να διεκπεραιώνονται και γρήγορα και να εκαθαρίζονται υποθέσεις κάποιων τραπεζών που δεν είναι βιώσιμες, ε, τότε παίζουμε με τη φωτιά. Το βλέπουμε ήδη και στην Ισπανία. Και δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω. Ε, στο CRD4 ε, κάντε πολύ στιβαρές και γερές προτάσεις γιατί εκεί θα μετρηθούμε όλοι και η αξιοπιστία της Ευρώπης που θέλουμε σήμερα να χτίσουμε. Αν θέλετε να έχετε και απαντήσεις, γιατί είναι πέντε οι συνάδελφοι, να είστε σύντομοι. Γιατί 6,5 ώρα τέλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη συνεργασία του και το πνεύμα συνεννόησης που δείχνει. Το σύστημα είναι πολύ ακριβό Τώρα στο θέμα της δανειοδότησης και της δανειοβλήψιας lending και borrowing. Υπάρχει μια πρόταση που εγώ είμαι εισηγητής για τα ενυπόθηκα ε, δάνεια. Γνωρίζει ο Επίτροπος ότι είναι ένα πρώτο βήμα και μόνο. Το δεύτερο, το country reporting. Ε, αυτό είναι μια δέσμευση ε, της Συμφωνίας Omnibus 2. Στο Στρασβούργο ε, κάναμε μια συνεδρίαση και ήταν ε, ευρία συνένεση του Κοινοβουλίου ότι θέλουμε οριζόντια ρύθμιση με διαφάνεια για την οδηγία, την 7 ε, για την ε, τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Και ο Επίτροπος Μπαρόσο, ο Πρόεδρος Μπαρόσο μάλιστα μιλάει για διαφάνεια. Υπάρχει οριστική απόφαση για αυτό το θέμα και ένα τελευταίο, ο διάλογος με τους χρήστες των χρηματοοικονομικών ε, υπηρεσιών. Για μας είναι πολύ σημαντικό, ε, αλλά πολλές φορές ε, οι χρήστες είναι οι προμηθευτές. Δεν είναι μόνο οι προμηθευτές της βιομηχανίας, αλλά είναι και τα μίντια, κυρίως ο τύπος που είναι δημόσια μέσα ενημέρωσης που ενημερώνει για το τι συμβαίνει ε, στις χρηματαγορές και γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι προμηθευτές της βιομηχανίας οι τράπεζες. Η κυρία Φερέιρα και άλλοι συνάδελφοι ακολουθούν ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Είμαι βέβαιη ότι και εσείς θέλετε να υπάρξει μια καλή διευθέτηση και καλή και σωστή επιτήρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ γιατί αναφέρατε τη σημασία των δοκιμών αντοχής και της επανικοδόμησης εμπιστοσύνης, όχι μεταξύ πολιτικών νομοθετών δηλαδή και των αγορών, αλλά και μεταξύ όλων των ανθρώπων που εκπροσωπούμε και των δημοτοπιστωτικών υπηρεσιών. Για μένα αυτές οι δοκιμές αντοχής είναι κάτι το ζωτικό. Έγιναν πέρυσι, θα γίνουν και φέτος. Στο περασμένο Στρασβούργο μερικοί από εμά, από την Επιτροπή μας, αγρύπνησαν για να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει με τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής και το ερώτημα που θέταμε όλοι ήταν γιατί τα κρατικά χρέη κρατιούνται από τα βιβλία των τραπεζών που δεν έχουν δείξει καμία, ε, κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ επίσης για αυτά που είπατε για, uh, για τη ρευστότητα πρέπει να υπάρχει ρευστότητα και μέτρα ρευστότητας για να έχουν ρευστότητα οι τράπεζες. Από μια χώρα που γνωρίζετε καλά ιδίως, μερικοί λένε ότι κάτι τέτοιο θα είχε πραγματικές θετικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων μονή μακρόπνων προγραμμάτων. Ότι δηλαδή αν οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα θα μπορούσε αυτό να ζημιώσει πραγματικά, να καταστρέψει το μέλλον της Ευρώπης και της οικονομίας της. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις είναι κάτι που απαιτεί ρευστότητα, το έχουν πει αυτό και οι ασφαλιστές. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε να πάρετε ως μέτρα για τις μακρόπνοες ή μακροχρόνιες επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με την ομιλία που μας στείλατε και από το Πανεπιστήμιο του Χάμπολτ, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε, όπως και γενικότερα, τη διάσταση των ε, πολιτικών της Ευρώπης σε αυτές τις τόσο δύσκολες, ταραγμένες στιγμές. Γι' αυτό έχω να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για κάποια άλματα που πρέπει να, γίνουμε, να γίνουν. Ομιλίες και κείμενα όπως αυτά θα πρέπει να ακούγονται και στο κολέγιο των επιτρόπων μιλήσατε στην ανάγκη να μιλήσουμε, ε, να δημιουργήσουμε ένα φόρο για την ε, φορολόγηση των εμπορικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μία ημερομηνία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει την επίτευξη του στόχου αυτού, Όπω και για τα ευρωομόλογα θα την έχουμε. Μπορούμε να υπολογίζουμε στη δική σα επιρροή στο Κολέγιο των Επιτρόπων ώστε να γίνουν κάποια άλματα πρόοδου, να ε, ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση για τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα. Το δεύτερο σημείο, το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με μια από τι επιτυχίε τη Επιτροπή και του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή το δημιούργημα ενό αρχιτεκτονήματο εποπτεία. Σε αυτό το αρχιτεκτόνημα σε αυτό το οικοδόμημα ενοσχύθηκε ο ρόλος των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Όμως το σημαντικότερο είναι στην πράξη και καθώς παράγονται νομοθετικά κείμενα, αυτό να, να, να μην υπονομεύει το κύρος και την λειτουργία των ευρωπαϊκών αρχών ακριβώς. Ήθελα λοιπόν συγκεκριμένα να ξέρω για το short selling και τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει η ΕΣΜΑ όπως προβλέπονται και εδώ στην ε, ε, έκθεση Καλφά που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και στην ε, θέση της Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες αυτές της ΕΣΜΑ που είναι θεμελιώδους σημασία, ώστε στο επίπεδο του short selling να μην υπάρξει κατακαιρματισμός των αγορών σε εθνικά επίπεδα. Μπορούμε εκεί να υπολογίζουμε στην ενεργό παρουσία και την επιρροή της ε, Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή. Και τρίτη παρατήρηση για την πρωτοβουλία που θα αναλυφθεί από το Σεπτέμβριο για την εξακολούθηση που αναφέρατε κι εσείς, ε, την εξακολούθηση που θα δοθεί στα θέματα αντιμετώπισης της κρίσης. Εδώ ε, να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Αυτά θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των τεστ κοπόσεως. Ε, όμως το Συμβούλιο στις 23 και 24 με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισε τελικά ποιο θα παρέμβει μετά τα τεστ κοπόσεων θα είναι, κοπόσεως θα είναι τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτό αντίκειται στις ε, διαθέσεις ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης που είχαμε εκφράσει με την έκθεση αυτή και που συμμεριζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την κρίση λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση δημιουργίας ε, ε, ε, ανέλυξης και περαιτέρω επιπλοκής με τα δημόσια χρέη και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Αυτό μας ανησυχεί, διότι χάνουμε κάπως το ρυθμό δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο. Με συγχωρείτε γιατί ξεπέρασα λίγο το χρόνο ομιλίας μου. Thank you very much, Mr. Commissioner. Ευχαριστώ Δύο ερωτήματα. Πρώτον, σαφώς είστε κάποιος που παίζει σημαντικό ρόλο, συνεννοείστε με όλους τους υπουργούς οικονομικών της Ευρώπης. Τι βλέπετε να τάση να παρατηρείτε μεταξύ τους. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να δαπανά περισσότερα από όσα κερδίζει ως έσοδα φορολογικά. Επομένω, το πρόβλημα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε τι οφείλεται. Δεύτερον, Ορισμένοι αναφέρθηκαν σε ακάλυπτα CDS. Κάποιος μίλησε για την ανάγκη εδώ η πλανή μου ε, μακροπρόθεσμων επενδύσεων αλλά και για υγιή διαχείριση των τραπεζών. Η απαγόρευση των ακάλυπτων δραστηριοτήτων ήταν ένας από τους λόγους μάλλον της κρίσης. Οι επενδυτικές τράπεζες ανέλαβαν αυτό το ρίσκο και όταν ακούτε ότι ίσως αυτό να επηρεάσει αρνητικά και τις σχέσεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα ή ότι δεν πρέπει να εγκρίνονται τέτοιες ακάλυπτες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν με κάποια συνέπεια παντού. Και εμείς ως νομοθέτες τι μπορούμε ακριβώς να κάνουμε για να το διασφαλίσουμε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λυπάμαι που δεν ήμουν από την αρχή στη συζήτηση. Ήμουν υποχρεωμένος να παρευρίσκομαι σε άλλη επιτροπή καθώς ήμουν εισηγητής. Άλλη ερώτηση είχα προετοιμάσει, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σύντομα επίγουσας, επίγουσας, ε, επίγοντο, ε, που έχει επίγοντα χαρακτήρα για τη χώρα. Όπως γνωρίζετε, χτες η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πουλάει άμεσα όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγημένες στο χρηματιστήριο και που έχει μερίδιο το δημόσιο. Ο κατάλογος μεγάλος. Είναι μια πολιτική που την οθείται εκποίησης δημόσιας περιουσίας και η Κομισιόν. Το ερώτημα που θέτω είναι, σε αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έχουν μετοχές μικροκαταθέτες και ασφαλιστικά ταμεία. Και το ερώτημα, ανεξάρτητα ποια είναι η άποψη του καθενός αν πρέπει να γίνουν ή όχι αυτές οι ιδιωτικοποίησεις, αυτή η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Θα επαναληφθεί το κακό προηγούμενο που έγινε με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα όπου κατά παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας όπως ενδεχομένως έχετε αφήσει να εννοηθεί είναι μια ερώτηση που σας έχω κάνει δεν έχω σαφή απάντηση όπου το πακέτο των μετοχών το πήρε η Deutsche Telekom χωρίς να γίνει δημόσιος διαγωνισμός. Και το ερώτημα είναι, κύριε Επίτροπε, εντάξει, γίνεται αυτή η διαδικασία. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα έχουμε παραβίαση, εν πάση περιπτώσει, της κοινοτικής νομοθεσίας για άλλη μια φορά, που σημαίνει μικρομέτοχοι και ασφαλιστικά ταμεία θα χάσουν χρήματα και όλη αυτή η υπόθεση θα χαρακτηριστεί ως κερδοσκοπικό πανηγύρι μεγάλων πολυεθνικών εταιριών γερμανικών κυρίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame Κύριε Μπέρες, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχω μια μικρή ερώτηση ενημερωτική. Μιλήσατε για τη Βασιλεία Τρία. Γνωρίζουμε όμως τώρα ότι η Βασιλεία 2 δεν εφαρμόζεται καλά. Δεν έχει μεταφερθεί μάλιστα σε κάποια κράτη-μέλη. Και τι προτίθεστε να κάνετε σχετικά με αυτό. Στη συνέχεια έχω δύο ερωτήσεις. Πιο τεχνικές. Είπατε σε σχέση με τα όσα είπε ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με την ανάγκη διοργάνωσης. Πώς τα λένε αυτά στα γαλλικά τώρα, δεν μου έρχεται. Το country reporting. Πώς το λένε αυτό. Παρουσίαση αναχώρα ε, των ισολογισμών των επιχειρήσεων, κυρίως των εξορρυκτικών που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην εκμετάλλευση ε, κάποιων αναπτυσσόμενων κρατών. Ωραία. Σε αυτό το πρόβλημα όμως το συγκεκριμένο τίθεται το εξή ερώτημα τα λογιστικά πρότυπα ποιος τα ορίζει. Και ε, η διακυβέρνηση του ERSB. Ο προκάτοχός σας είχε ρίσει μια ομάδα παρακολούθησης, monitoring, για αυτορύθμιση και αυτοεποπτεία παρακαλώ. Ε, πέρα λοιπόν από τα συγκεκριμένα πρότυπα αναχώρα, τι θα κάνετε εσείς για το θέμα αυτό πολύ δε περισσότερο που αν θέλετε να ενδιαφερθείτε και να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να συνεργαστείτε με τον συνάδελφό σας κύριο Σεμετά για να δείτε τι θα γίνει από πλευράς φορολογίας. Ένα τελευταίο και το σημαντικότερο σου ερώτημα. Όλη η με αυτή για την οποία έχετε εργαστεί πολύ εσείς ε, ε, με σκοπό να δημιουργηθούν κάποιοι θεσμοί για τη σταθερότητα των χρηματαγορών. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι κάθε κίνηση κεφαλαίου δεν είναι κατά ανάγκη προστιθέμενη αξία για την οικονομία που τη δέχεται αυτή τη συναλλαγή. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί σήμερα ανησυχούν για αυτά τα φαινόμενα και βλέπουμε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικές φούσκες είτε πρόκειται για τον τομέα το κατασκευαστικό της οικοδομής ή για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες που πέφτουν όμοιροι, ε, ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ κρίσιμες μακροοικονομικές καταστάσεις. Ξέρω ότι ένας επίτροπος δεν μπορεί άμεσα να επέμβει για να ε, καταρτήσει μια οδηγία. Αυτή η πρόκληση όμως είναι υπαρκτή. Εσείς πώς σκέφτεστε να ανταποκριθείτε, να αντιδράσετε. Και ένα τελευταίο. Αν θέλουμε να έχουμε μέσα εργαλεία στη διάθεσή μας για να δούμε τι γίνεται ε, και πώς λειτουργούν οι ε, χρηματαγορές, ξέρω ότι στην Κεντρική Τράπεζα ορισμένοι ανησυχούν για την τίτλοποίηση, για τους τίτλους μάλλον, η ενημέρωση για τους τίτλους να θεωρείται δημόσιο αγαθό. Γνωρίζετε ότι ο συνάδελφός σας που έχει ως χατοφυλάκιο τον ε, ανταγωνισμό ε, μίλησε με ανησυχία για τη Standard Poor's που ε, πουλάει κάποιες προφορίες οι οποίες κανονικά θα πρέπει να είναι δημόσιες. Και μια που είστε αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα για τις αγορές αυτά τα θέματα πρέπει να σας ενδιαφέρουν και να σας... Ορίστε κύριε Επίτροπε, αυτά τα ολίγα, λέει η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Έχετε μέχρι 20 το χρόνο να απαντήσετε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τους διερμηνείς για την υπέρβαση ωραρίου. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και συνεκτικός, αλλιώς θα συμπληρώσω γραπτός τις απαντήσεις μου γιατί έχω και εγώ κάποιε ανηλυμένε χρεώσει Ήδη θα έπρεπε να είχα αναχωρήσει για άλλη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Η κυρία Μακάρθη ε, ε, ανέκαμψε και ευχαριστώ για την παρουσία σα. Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα και εγώ δεν πιστεύω στην αυτορύθμιση. Ήταν πολύ μεγάλη επίβολη ιδέα, όσο και κακή όμως στην αρχή της παγκοσμιοποίησης των συναλλαγών θεωρήσαμε ότι οι αγορές θα αυτορυθμίζονται και ότι ε, οι ελεύθερες συναλλαγές θα μπορούσαν ε, να ρυθμίσουν τα πάντα χωρίς κανόνες και χωρίς διακυβέρνηση. Ξέρουμε ότι είναι μύθος αυτά. Και εβδομάδα, τη βδομάδα βλέπουμε στο G20 με ποιο τρόπο προσπαθούμε να στήσουμε πλέον μια παγκόσμια διακυβέρνηση, στο εσωτερικό της οποίας θα πρέπει να ευρεωθεί η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η κυρία Μακάρθη με ρώτησε και για την τραπεζική κρίση στην Ιρλανδία. Σημειώνω ότι οι κραδασμοί που έχουν πλήξει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία δεν είναι όλοι της ίδιας φύσεως. Η κυρία Μακάρθη, το έχω ξαναπεί και το πιστεύω. Πριν από δύο χρόνια, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, ας πούμε, και των Ιρλανδικών τραπεζών, Αν είχαμε τα εργαλεία και τα άλλα μέσα πρόνοιας, εποπτείας και επίλυσης αυτών των θεμάτων, εξωτερικής και εσωτερικής, αν όλα αυτά τα εφαρμόζαμε σωστά και είχαν στηθεί ήδη από τότε, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η κρίση αυτή των τραπεζών θα ήταν πολύ πιο ήπια ορισμένα προβλήματα, συγκρούσεις συμφερόντων, διαπλοκή στα συμβούλια, τα διοικητικά, η αποτυχία δυναμίες της εποπτείας άφησαν να δίνουν έτσι άκρητα δάνεια ε, με τρόπο πάρα πολύ γενναιόδωρο και ανεξέλεγκτο. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εάν τα μέσα και τα εργαλεία που σήμερα επεξεργαζόμαστε από πλευράς εξωτερικής και εσωτερικής εποπτείας, επίλυσης και διακυβέρνησης τα είχαμε τότε. Γι' αυτό άλλωστε κυρίες και κύριοι λέγω και πάλι ότι χρειάζεται σοβαρή δουλειά αλλά και ταχεία γιατί οι αγορές και τα προβλήματα καλπάζουν. Έχουν άλλους χρόνους, πολύ πιο γρήγορους από τους χρόνους της δημοκρατίας. Βεβαίως θέλω πάντα να σας ε, ενημερώνω με ακρίβεια για ε, τις ε, διατλαντικές συνεννοήσεις. Για τρίτη φορά θα πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες την άλλη εβδομάδα και να συναντηθώ με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, τις ρυθμιστικές αρχές, αποπτικές αρχές και στα πλαίσια του G20 ε, να δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες και θα έρθω να συμπληρώσω αυτά τα στοιχεία ε, από την Κίνα και τις άλλες χώρες. Προς το παρόν οι συναλλαγές είναι κατά 80% διατλαντικές, δηλαδή Ευρώπη-Αμερική. θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ για τον ε, τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία εκεί και απαντώ και στην κυρία Μπερές εδώ για το ΙΑΣΠ ε, τι ε, μπορεί να γίνει ως προς τη σύγκληση των λογιστικών προτύπων Αυτές οι ιστορίες fair value, market value, ποια είναι η αγοραία αξία, η δίκαιη αξία, δεν είναι πάντα θέμα συζήτηση μπορεί να είναι και θέμα διαφωνίας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών. Πραγματικά πιστέψτε με, ασχολούμαι σε λεπτομέρειες με αυτά τα θέματα και σε σχέση με τους Αμερικανούς και σε άλλα θέματα που δεν ε, είναι αμέσως αρμοδιότητα της δικής επιτροπής όπως είναι τα δημόσια έργα. βλέπω μια πολύ μεγάλη ανισορροπία σε ό,τι αφορά την διάνοιξη των δικών μας αγορών σε αμερικανικές εταιρείες χωρίς να υπάρχει αμοιβαιότητα. Χρειάζεται όμως να ε, εφαρμοστεί ε, η ε, συμφωνία GPA που δεν έχει εφαρμοστεί ως ε, όφιλε. Θα σας αναφέρω κυρία Πρόεδρε και σε εσά και στα μέλη της Επιτροπής σας μετά την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ και το CRD3 που γνωρίζετε πολύ καλά κυρία Μακάρθη Και πάλι παρακολουθούμε πολύ στενά αυτά τα πράγματα. 15 κράτη-μέλη σήμερα έχουν κοινοποιήσει επιπλέον μέτρα ε, μεταφοράς. 6 κράτη αναφέρουν ε, μερική μεταφορά στην νομοθεσία και ε, άλλα έξι δεν μας έχουν κοινοποιήσει τίποτα και κινητοποιούμε τις διαδικασίες προσφυγής επί παραβάση για τα τελευταία αυτά έξι κράτη. Το πιο καθόδες θέμα είναι ποια είναι η δική μας τώρα αξιολόγηση, κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες ε, της οδηγίας αυτής. Τα κράτη-μέλη που έχουν μεταφέρει στην ομοθεσία τους το πράτών σωστά και οι τράπεζες ε, τα εφαρμόζουν ορθά. Εγώ δεν είμαι υπόπτης των τραπεζών και των κρατών. Ε, είμαι υποχρεωμένος να εμπιστεύομαι τις κρατικές εποπτικές αρχές για το ότι εφαρμόζεται σωστά το CRD3 ε, και οι τράπεζες κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Κυρία Μακάρθη, θα υπάρξει και ένα κοινό εργαστήριο workshop ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το βλέπω θετικά. Και σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, συμπληρώνω την απάντησή μου λέγοντα ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε τι μεταρρυθμίσει που τρέχουν αυτόν τον καιρό. Οι Ιρλανδικέ αρχέ κάνουν ε, ένα πολύ δύσκολο έργο, πολύ θεραλέο και ε, εμπιστευόμαστε και το πρόγραμμα στήριξης ε, της Τρόικα στην Ιρλανδία. Κύριε Γκίγκολτ, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας από πολλά θέματα και την επαγρύπνησή σας. Πρέπει να σας πω ότι ε, σε όλους αυτούς τους κραδασμούς πάντα που πλήττουν την Ελλάδα, την Ελλανδία, την Πορτογαλία ενδεχομένω και άλλες χώρες, είναι πολλά τα στοιχεία. Μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι πολλές κρίσεις μέσα στην κρίση. Γι' αυτό έχουμε τόσο βαριά ευθύνη αυτό τον καιρό. Και γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε πολύ την ψυχραιμία μας και με μια αλληλεγγύη. Θέλω να σας πω εγώ την πεποίθησή μου. Γι' αυτό απέτησα και φοροτιμή στην εργασία του ΟΛΗΡΕΝ. Θα μπορούσα όμως να αναφέρω και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλές κυβερνήσεις. Απέναντι στις κρίσεις αυτές τους κραδασμούς, που δεν πλήττουν μόνο την Ευρωζώνη, την Ευρωζώνη ως ζώνη, αλλά τα κράτη της Ευρωζώνης, έχουμε προχωρήσει. Επιτέλους, Έχουμε κάποια στοιχεία διακυβέρνηση και θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να φροντίζουμε, να τα εφαρμόσουμε για την Ευρωζώνη, για την ευρωπαϊκή οικονομία που κανονικά θα έπρεπε να ε, τα είχαμε θεσπίσει πριν από 10 χρόνια. Και το λέω εδώ μπροστά στην κυρία Μπερέ, στη συντακτική συνέλευση. Ήταν και η ίδια πρόεδρο σε μια ομάδα εργασία για την οικονομική διακυβέρνηση. Και το θυμάστε ίδια. Ότι ε, ήταν Σηγεί ηχθείω. όχι, όχι οι εργασίες της Επιτροπής, τα αποτελέσματα. Ε, μπορεί να το πει και ο κύριος Μένες Δεβίγο, ήταν και αυτός παρόν. Και δεν ήταν πριν από 10-15 χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια. Τώρα κάνουμε αυτά που έπρεπε να είχαμε κάνει όταν ε, ήρθε το ευρώ. Ε, η εποπτεία στον προϋπολογισμό, η αλληλεγγύη στα οικονομικά κτλ. Αυτό που ισχύει κύριε Γκίγκολτ, το είπα άλλωστε και στο Βερολίνο της προάλλες, είναι το εξή. Καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν είναι μόνη της, αλλά και καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι απαλλάσσεται από την τήρηση της πειθαρχία που συμφώνησε με άλλους αυτόν τον εσωτερικό κανονισμό της κοινή μας ε, ε, ιδιοκτησίας που είναι η Ευρωζώνη. Και βεβαίω χρειάζονται κανόνε και για διαφάνεια και για διοντολογία και για ε, ηθική. Θα πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα καθήκοντά τη στη χώρα τη. Εσεί προέρχεστε από μια χώρα, κύριε Γκίγκολτ, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ανεξάρτητα από του κυβερνητικού ε, σχηματισμού ή συνασπισμού, έχει μια κουλτούρα τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δηλαδή, η ανάπτυξη σταθεροτητα δηλαδη η αναπτυξη οικονομια δεν μπορεί να οικοδομηθεί ε, πάνω σε δάνεια, ε, δηλαδή με ε, ακάλυπτες επιταγές που μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενναίες και πολλές φορές το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα που εξάγουμε από την κρίση αυτή. Πάντως γίνεται πρόοδος και στην διακυβέρνηση, την οικονομική και στην Ευρωζώνη. Κύριε Γκίγολτ, αρχάς Ιουλίου θα δημοσιεύσουμε το κείμενό μας για το CRD 4. Σας ακούω και πάλι. Έχουμε και φιλοδοξίες. Θέλουμε να εφαρμοστεί η Βασιλεία 3. Επίσης, η Επιτροπή της Βασιλείας ίδια θέλω ε, να ελέγξω κατά πόσο είναι σίγουρη για τα όσα προτείνει. Παράδειγμα, για τη ρευστότητα γνωρίζω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες, διότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο. Για τους δείκτες μόχλευσης, leverage ratio, σύμφωνα με τους αρμόδιους και τους κεντρικούς τραπεζίτες αυτό θα είναι πρώτα στο δεύτερο πυλώνα με μια περίοδο παρατήρησης ε, πολλών ετών μέχρι το 2016 συγγνώμη, και δεν θα το προτείνουμε ως μέτρο του πρώτου πυλώνα γιατί δεν είναι αρκετή ευκρίνεια και ακρίβεια για την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες που θα έχει ως δεσμευτικό μέσο. Κύριε Γκίγκολ, θα πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου και θα το πράξω και πρέπει να προσέχω. Και εσείς ο ίδιος μιλήσατε για χρηματοδότηση. Πώς το είπατε. Όχι εσείς κάποιος άλλος συνάδελφος. Η κυρία Φόρτ. Ναι, μισό λεπτό. Νόμιζω η κυρία Φόρτ, είπε και ο κύριο ε, Καμάλ, για τις μακροπρόθεσμες ε, χρηματοδοτήσεις λοιπόν, θα πρέπει εγώ να προσέχω να ε, παρακολουθώ τι γίνεται στι ευρωπαϊκές οικονομίες και τι συνέπειες. Καλέ οι εκκλήσει στις τράπεζες ή προειδοποιήσεις των τραπεζών, ε, αυτά δεν με εντυπωσιάζουν, ξέρετε. Τα ακούω, τα σημειώνω, όπω ακούω όλε τι κυβερνήσεις που εκφράζονται σχετικά. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και ε, του χώρου που καταλαμβάνει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κύριος Σάντς Πρεσέδο μίλησε για τα ενυπόθηκα δάνεια και που είναι ο ίδιος ε, εισηγητής. Είναι μια πρώτη φάση μόνο και ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Το πεδίο εφαρμογή θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε τρία χρόνια, αλλά καλό θα είναι να αρχίσουμε από την καταναλωτική πίστη. Και εσεί, κύριε σας Πρεσέδο, όπως και η κυρία ε, ε Μπερές αναφερθήκατε στην αφορά αναχώρα, country by country reporting. Σας είπα είναι προτεραιότητα για μα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής τη αναδυόμενε οικονομίε ιδιαίτερα τη Αφρική, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επ' αυτού. Τώρα το ιδεώδες θα ήταν να υπάρξει ένας παγκόσμιος συνολικός συντονισμός και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε κυρία Μπερές στα πλαίσια του EASB. Προσωπικά συμμετέχω ε, με μεγάλη φροντίδα σε όλες τις συνεδριάσεις του EASB. Δεν έχω χάσει καμία. Στις 13 Ιουλίου θα μεταβώ στην Νέα Υόρκη για την επόμενη και θα είμαι παρόν σε όλες τις συνεδρίες, Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, άλλωστε είναι συναρπαστική η εργασία εκεί. Και μάλιστα με τον εκλειπώντα κύριο Παντό Σκιάπα εργαζόμαστε εκεί για μεγαλύτερη διαφάνεια, για μεγαλύτερο σεβασμό του monitoring board από τους trustees και εργαζόμαστε ακριβώς για μεγαλύτερη διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς και όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού και μετά από συνεννόηση των ε, μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, του οποίου είμαι μέλος. Πέρα όμως από τη διακυβέρνηση αυτή governance και τη καλύτερη συνεννόηση των διαφόρων ε, φορέων, θα δω και τις λεπτομέρειες για ε, τα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται εκεί. Βέβαια έχω εκφράσει και ανησυχίε, ξέρετε, για το leasing και για άλλα θέματα πρόσφατα. Επαναλαμβάνω και στον κύριο Σάντσες Πρισέδο και στην κυρία Μπερές ότι αυτό το όργανο είναι όργανο σύγκλησης. Δεν θα πρέπει να καταλήξει στο αντίθετο. Εργάζομαι προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς καμία εμ, αφέλεια ή η υπόθεση αυτή του country by country reporting δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιμένει τι θα βγει από εκεί. Ε, θα πρέπει και η ίδια να δείξει ηγετική στάση. Ε, αρχές 2011 ε, κάναμε μία έρευνα. Ε, έχουμε λάβει αποφάση, απαντήσεις συγγνώμη, πάνω από 80 ο κύριος Μπαρόσο προτιμάει την οδηγία για τη διαφάνεια για ένα πολύ απλό λόγο, αντικειμενικό, γιατί θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο και αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Όμως, το είπε και ο κύριος Γκίγκολτ και η κυρία Μπερέ, πιστεύω, έχουμε και την οδηγία για τα λογιστικά πρότυπα που αναθεωρείται και θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη το Σώμα των Επιτρόπων το συζητούμε και αφού σας άκουσα με μεγάλη προσοχή θα το ε, διαβιβάσω εκεί και θα το προωθήσω με σθένος και με πειθό, αλλά χρειάζεται κάποια εργασία και κάτι άλλο και παρακαλώ να με καταλάβει. Το πεδίο εφαρμογή επίσης αυτής της μελλοντικής νομοθεσίας μας απασχολεί θα είναι μόνο εξορρεκτική βιομηχανία που είναι πάρα πολύ ισχυρή και σημαντική, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς, όχι μόνο αυτοί, που εγώ είμαι υπέρ, ας πούμε, τι γίνεται ε, με την υλοτομία, γενικά την εκμετάλλευση των δασών. Και ε, απαιτήσει ε, τη διαφάνεια θα είναι αναχώρα, αναέργο. Θα πρέπει και αυτό να το κοιτάξουμε και να δούμε και το κόστος όλων αυτών των μέτρων που προτείνουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ δεν θέλω η Ευρώπη να έχει μικρότερη ε, ε, φιλοδοξία από ότι οι Αμερικανοί. Stress τεστ. Ο κύριος Κίγκολ και η κυρία Σουίμπρον το είπε και η κυρία Βίκη Φόρτ. Αυτό το καιρό διεξάγονται αυτές οι δοκιμές και είναι ε, πολύ πιο αυστηρές από τις προηγούμενες. Έχουμε ένα σενάριο συγκριτικά και αναλογικά δυσμενέστερο. Μεγαλύτερο έλεγχο των αποτελεσμάτων, πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιοποίηση και για το κεφάλαιο αναφορά και το benchmark. Όλα αυτά είναι πολύ πιο αυστηρά οι βάσει επίση και η κυρία Φερέιρα το είπε. Αυτές οι δοκιμέ αντοχής λοιπόν σε ε, ακραίες καταστάσεις θα μας βοηθήσουν για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και τα μέτρα που θα λάβουμε τώρα, το επόμενο backstop που εξαρτάται από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του. Και η προετοιμασία δεν θα πρέπει να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει ήδη από τώρα να εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Γκίγκολτ επίσης και η κυρία Φόρτ μίλησαν για το δημόσιο χρέος στο banking book Εγώ εμπιστεύομαι ε, τις επιλογές ε, ε, της τράπεζας του Λονδίνου που επέλεξε αυτά τα τεστ και αυτό είναι πρόοδος. Επίσης κυρία Φόρτ παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τι γίνεται με τα συνταξιωτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι το ίδιο κείμενο με τη Βασιλεία 3 για τη Βασιλεία 3 θα πρέπει να προετοιμάσω 600 σελίδες σχέδιο οδηγίας πλήρες, γιατί η φερεγγιότητα ε, μπορεί να είναι πολλές σελίδες τεχνικά ε, μέτρα. Πάντως, κυρία Φόρτ, πραγματικά για την ε, υπόθεση των ασφαλιστικών εταιριών και των συνδεξιδικών ταμείων το παρακολουθώ. Ναι, κυρία Φερέρα. Είμαι πολύ αποφασισμένος στο Σώμα των Επιτρόπων να ε, υποστηρίξω τα ομόλογα έργων, ε, project ε, bonds και ο κύριος Μπαρόσο και πολύ νωρί το είπα εγώ από την πρώτη τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής από τη στιγμή που διοριστήκαμε μίλησα υπέρ ενός φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και πρέπει να σας πω σε όλες τις συνεννοήσεις και επαφές που είχαμε με το Συμβούλιο και τούτη εδώ την εβδομάδα για τις ακάλυπτες πωλήσει, το short selling εγώ αγωνίζομαι να διαφυλάξω αυτά που λέει ο κανονισμός και με τη δική σας υποστήριξη. Και λέω στο Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να ξυλώσουμε ε, τα όσα έχουμε γράψει για την ΕΣΜΑ ως εξουσία στον κανονισμό. Και επίσης, καλό είναι να περιμένουμε και κυρία Φερέρα τα αποτελέσματα των stress test για να ε, προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση. Απάντησα προηγουμένως στον κύριο Καμάλ και στον κύριο Γκίγκολτ για τον τρόπο με τον οποίο οικοδομεί κάνει αηφόρο ανάπτυξη και λέω, επαναλαμβάνω, αυτό δεν μπορεί να γίνει με δάνεια και ε, Δαπανώντα πολύ περισσότερο από τα έσοδα που έχουμε. Για το short selling, το είπατε και εσείς κύριε Καμάλ, και τι συνέπειε έχει αυτό για τη ρευστότητα, είχα πάρει μια απόφαση στην αρχική πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προτείνουμε ε, την απαγόρευση των naked short selling, τις ε, ακάλυπτες πωλήσει για τα CDS, αλλά να αποφασίζουμε γρήγορα και από κοινού απαγόρευση όταν η κατάσταση στις αγορές το απαιτεί. Γρήγορα και από κοινού, όχι γενική απαγόρευση. Ε, αυτό είναι άλλωστε η πρόοδος του κειμένου για τις ακάλυψεις πωλήσει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Και απαντώ και στην κυρία Φόρτ για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Για μένα είναι προτεραιότητα. Έτσι θα έχουμε καλύτερη προσαρμογή και στο ΣΕΡΔΕΚ 4 και θα εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτή για να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλύτερα και επίσης συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ταγιάννη για την αύξηση των μέσων ή ε, την υποστηρίξη του κεφαλαίου κινδύνου, που είναι και αυτός ένας τρόπος υποστηρίξης των μακροχρόνιων επενδύσεων. Ο κύριος Χουντής ε, ανέφερε τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και φυσικά μπορώ να κατανοήσω πολύ καλά την ανησυχία σας κύριε Χουντή Λέω μόνο χωρίς να αναμειχθώ σε αποφάσεις που παίρνουν ελληνικές αρχές. Γνωρίζουμε όμως ότι το πράττουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο ε, με τη συμφωνία και το συμβόλαιο που έχουν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας διαβεβαιώ κύριε Χουντή ότι από τη θέση που βρίσκομαι θα φροντίσω το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο να γίνεται σεβαστό και ε, τη στιγμή των ιδιωτικοποιήσεων. Ε, σημείωσα αυτά που είπατε κύριε Μπερές για τη χρήση των πληροφοριών, τη χρηστή ε, διαχείριση από όλους τους φορείς, ε, τους χρηματοοικονομικούς. Ο κύριος Σαλμούνια, ξέρετε τι έκανε. Έχει τα μέσα αυτά στη διάθεσή του, θα το κοιτάξω κι εγώ, θα σας απαντήσω γραπτός γιατί πρέπει να μελετήσω τις προτάσεις σας και επίση, ο κύριος Σαλμούνια, ιδιαίτερα για το CDS έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για τον ανταγωνισμό. Αυτά. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ αγαπητέ Μισελ. Ε, στο επανειδήν θέλω να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που επέτρεψαν στον Επίτροπο να ε, ολοκληρώσει την τοποθέτησή του με τέτοιες λεπτομέρειες. Επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, δυστυχώς Δευτέρα 6 Ιουνίου, κανονικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ε, στο Στρασβούργο δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Τι να κάνουμε, 6 Ιουνίου επόμενη συνεδρίαση, λήξη.